Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επίτροπε, αγαπητέ Γενική Γραμματέα, αγαπητοί όλα, αγαπητοί Σουζάνε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους θερμά και να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Αντιπρόεδρος Αρμόδιος και μάλιστα με πάθος αρμόδιος για την πρόθεση της πολυγλωσίας στο θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα όργανο που η πολυγλωσία είναι νευραλγικό σημείο της ίδιας της ύπαρξης αλλά και της λειτουργίας αυτού του οργάνου. Θα ήθελα να ακούσω την αγαπητή ε, φίλη και επίτροπο Ανδρούλα Βασιλείου αρμόδια για την νεολαία, τον πολιτισμό, την παιδεία και την πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης θα ήθελα να ακούσω και να ε, καλωσορίσω για την παρουσία του τον Κλάους Βέλε που είναι ε, ε, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους μας. Όπως ξέρετε, σήμερα ξεκινά η διάσκεψη κορυφής η... το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γι' αυτό θα ήθελα τη δική μου παρουσίαση να την περιορίσω σε ένα θερμό χαιρετισμό και αφού ακούσουμε ε, τους ε, ομιλητές μας, τους καλεσμένους μας, θα επισέλθουμε ε, στην ουσία όπως αυθόρμητα θα ήθελα να κάνω σε ένα τόσο σημαντικό και κορυφαίο ακροατήριο. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η συνάντηση, εξαιρετικά σημαντική, γιατί εκπροσωπούνται εδώ πάρα πολλά θεσμικά όργανα, ιδρύματα, οργανώσεις και είναι και κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων αυτών των οργάνων. Γι' αυτό και η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια εκδήλωση και πρωτοβουλία που αν θυμάμαι καλά είναι άνευ προηγουμένου. Είναι πραγματικά προδότυπη και από την οποία περιμένουμε πάρα πολλά. Γιατί εδώ έχουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά να πούν και έχουν τεράστια προσφορά στον τομέα της πολυγλωσίας Έχουμε πολιτικούς ε, φορείς ε, από τα θεσμικά όργανα, Βρυτάνης από πανεπιστήμια και ηθήνοντες για την ε, επιμόρφωση των ε, διερμηνέων συνεδρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες χώρες, από Λίβανο, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και από μερικές χώρες της Αφρικανικής Επίρου. Έχουμε επικεφαλής των υπηρεσιών διερμηνίας ε, εθνικών και διεθνών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στη ΧΙΝΤΣ και επίσης έχουμε και μέλη της ΕΙΣΤΗ και και την, της IAML-ADP. Επίσης έχουμε και εκπροσώπους ε, ερευνητών στον πολύ σημαντικό τομέα των νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστώ θερμά την Γενική Διευθύντρια της Διερμηνίας, ε, την κυρία Όλγα Κοσμίδου, τη φίλη Όλγα Κοσμίδου, που αναφυσβήτητα είναι το Άγιο Πνεύμα και ξέρετε ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν αρμόδιο για την επιφύτηση ε, στις ε, γλώσσες, στην ε, μυθολογία τη χριστιανική. Και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο και με αυτή την ιδιότητα έχει διοργανώσει αυτή την διάσκεψη η Όλγα και φυσικά θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε θερμά και να εξάρουμε την συμβολή της. Επίσης, θα ήθελα να κάνω και κάποιες σχέσεις ε, αργότερα και προσωπικέ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Βασιλείου, τονίζοντα ότι μόλις επέστρεψα από την πατρίδα της ε, και θα ήθελα να εξάρω το κορυφαίο έργο της Κυπριακής Προεδρίας κατά το εξάμεινο της Κυπριακής προεδρία Με ιδιαίτερη χαρά αναγνωρίζω το έργο σας αγαπητή Ανδρούλα, γιατί πραγματικά είστε υπόδειγμα και για θέματα σχέσεων μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ευχαριστώ θερμά, Ανδρούλα, και έχεις το λόγο. Dear friend, Vice President. Ε, Αγαπητοί φίλοι, Αντιπρόεδρε, Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Κοσμίδου, αγαπητοί Πριτάνης, είναι μεγάλη μου χαρά να κάνω την ε, εισαγωγική ομιλία στη σημερινή διάσκεψη και αυτό με χαροποιεί ακόμα ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα είχε γίνει και η ακρόασή μου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να διοριστώ ως Επίτροπος. Η πολυγλωσία ε, ήταν στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή, τη δεκαετία του 50. Η εκμάθηση γλωσσών βοηθά όλους τους πολίτες να ανθίσουν πολιτιστικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Ανοίγει το μυαλό των ανθρώπων στην υπέροχη πολυμορφία που είναι τόσο ουσιαστική για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Γι' αυτό μια από τις προτεραιότητες μου ως Επιτρόπο είναι να στηρίξω όχι μόνο τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης τις 60 περίπου ευρωπαϊκές γλώσσες μειονότητας ή περιφερειακές γλώσσες. Επίσης πιστεύω πω πρέπει να προωθηθεί η εκμάθηση των γλωσσών από νεαρή ηλικία. Πριν από 10 χρόνια στη Βαρκελόνη οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισαν ε, ένα φιλόδοξο όραμα για την εκμάθηση γλωσσών και τη συμβολή της, ε, τη συμβολή της εκμάθησης γλωσσών σε κάθε, για κάθε παιδί και την εκπαίδευσή του η βελτίωση των βασικών ε, δεξιοτήτων κυρίως μέσω της ε, διδαχής δυο άλλων γλωσσών πέρα από τη μητρική γλώσσα, η πρώτη γλώσσα του κάθε παιδιού από πολύ νεαρή ηλικία. Σήμερα είναι φυσιολογικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε πόσο χρήσιμο ήταν αυτός ο στόχος της Βαρκελόνης, πόση πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, ποιος ήταν ο επόμενος στόχος παρά τη βαθιά οικονομική κρίση, η πιο, ο πιο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αλλάξει. Συνεργασία για μια καλύτερη κοινωνία με πλήρη σεβασμό στις διαφορές μας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως η ελευθερία, η ισότητα, η ελληνική και η διαφορετικότητα μπορούν να συνδυαστούν σε μια κοινή προσπάθεια και η γλώσσα είναι ουσιαστική για αυτή την εκπλήρωση αυτή της αποστολή. Ω επίτροπο υπεύθυνη για την παιδεία, τον πολιτισμό, την πολυγλωσία και την νεότητα, προσδίδω μεγάλη σημασία στη συμβολή των ε, δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλλουν στον τομέα των γλωσσών ε, και στην κοινωνία γενικότερα. Και γι' αυτό πιστεύω πως ε, σε έναν πιο κινητικό και διασυνδεδεμένο κόσμο η πολυγλωσσία έχει, αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα και αυτό δεν μπορεί να το αγνοεί κανείς. Σήμερα μιλάμε για τις νέες τεχνολογίες, την παιδεία και άμεσα η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης έρχεται στο μυαλό. Είναι αυτό ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίε διερμηνία τη Ένωση αλλά είναι και περισσότερο ώστε να στηρίξουν την κατάρτιση νέων διερμηνέων συνεδρίων σε ε, πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Νέε δε ευκαιρίε έχουν δημιουργηθεί μέσω δύο νέων καινοτομιών. Η πρώτη είναι το Αρχείο Ομιλιών που ξεκίνησε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και την Αρμόδια Διεύθυνση Διερμηνίας και που χρησιμοποιείται από φοιτητέ κυρίως για να ε, ασκηθούν σε σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Το Αρχείο Ομιλιών αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάνω από 2.250 βίντεο ταινίες που είναι διδακτικού περιεχομένου, πραγματικές ομιλίες για τη χρήση όλων των ευρωπαϊκών επισήμων γλωσσών, καθώς και κάποιων γλωσσών τρίτων χωρών. Αυτό το υλικό βοηθά τους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλώσσες τους, να ασκηθούν στις ε, δεξιότητες διερμηνίας. Δεύτερη σημαντική καινοτομία είναι οι διμερείς και πολυμερείς ε, εικονικές ε, διδασκαλίες. Πρόκειται για τηλεδιασκέψεις που συνδέουν ε, διερμηνείς από την Υπηρεσία δερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν με 15 ε, πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτών των εικονικών μαθημάτων ε, αξιολογούνται οι φοιτητές από επαγγελματίες δερμηνείς από τις Βρυξέλλες με βάση τις προδιαγραφέ που απαιτούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η ηλεκτρονική εκμάθηση βοηθά επίσης το προσωπικό της ίδιας της διεύθυνσης διερμηνίας, διερμηνής που μπορεί να βρουν ειδικευμένε γνώσεις για θέματα που συζητώνται στις συνεδριάσεις χάρη σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο. Και αυτό φυσικά αυξάνει την ποιότητα της ερμηνείας που παρέχουν οι διερμηνείς μας. την ε, διαδικτυακή πύλη κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από, για διάφορες διασκέψεις που διοργανώνονται από τις μονάδες διερμηνίας. Οι διαλέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ε, υλικό εκπαίδευσης, ε, άσκησης για τους συναδέλφους. Μια μεγάλη πρόκληση σε σχέση με τις τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διερμηνία είναι πρόσφατη και έχει έρθει στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, του ηφαιστείου του 2010. Εφόσον τα αεροπορικά ταξίδια ήταν πολύ περιορισμένα τότε, ε, χρειαζόταν να βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος για να συνδεθούμε με μακρινές ε, τοποθεσίες μέσω ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης με διερμηνία. Θυμάμαι πως ε, οι υπηρεσίε δερμηνίας της Κομισιόν κατάφεραν να διοργανώσουν ε, πολύ γρήγορα μια επίγουσα συνεδρίαση του, των επιτρόπων με διερμηνία για όλους, ακόμα και αυτούς που βρίσκονταν στις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες. Οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί έκτοτε, εν μέρη λόγω των αυξανόμενων περιβαλλοντικών προβληματισμών όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια και την μείωση των διοικητικών προπολογισμών και στα δύο ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη, αλλά επίσης λόγω των ευκαιριών που έχουν δημιουργηθεί χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη. Εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή βλέπουν καθημερινά πώς τα τηλέφωνά τους και οι ταμπλέτες κάνουν τη ζωή την καθημερινή ευκολότερη. Φυσικά αυτό αυξάνει τις προσδοκίες ε, σχετικά με το ποιες παρόμοιες τεχνολογίες, μάλλον τι μπορούν να επιτύχουν παρόμοιες τεχνολογίες σε επαγγελματικό πλαίσιο. Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτές τις τεχνολογίες θα είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε ε, πολύγλωση επικοινωνία υψηλού επίπεδου που βοηθάει και στηρίζει την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Μια κρίσιμη πτυχή της τεχνολογικής εξέλιξη είναι επίσης η χρήση των κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook και το YouTube. Οι υπηρεσίε δερμηνία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων γρήγορα αναγνώρισαν τις ευκαιρίες επικοινωνίας που προσφέρουν αυτά τα μέσα και τα χρησιμοποιούν εκτεταμένα ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στους νέους για να τους προσελκύσουν στο επάγγελμα του διερμηνέα. Το να αντισταθεί κανείς στις τεχνολογικές αλλαγές είναι αδύνατον. Η τεχνολογία έχει ανατρέψει την κοινωνία σε πολλές, πολλές περιοχές ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, νέα είδος ε, εκμάθησης των γλωσσών έχει προκύψει. Το ίντερνετ αποτελεί ένα μέσο μέσα από το οποίο ο κόσμος μπορεί να μάθει, να μοιραστεί και να συνεργαστεί με τρόπους που παλιότερα δεν μπορούσαμε να το, να το φανταστούμε. Ωστόσο, η διαρκής επιτυχία προέρχεται από την προετοιμασία των φοιτητών για την αλληλεπίδραση και την εκμάθηση από όλα αυτά τα νέα περιβάλλοντα. Και γι' αυτό και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να έχουμε σύντομα αποφύτους με το σωστό μείγμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Φυσικά είναι καλό να ενσωματωθεί η χρήση της τεχνολογίας στο βασική εκμάθηση γλωσσών, αλλά πρέπει να μπορούμε να δείξουμε ότι καθιστά την διδασκαλία πιο αποτελεσματική. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιδιώκουμε τη χρήση τεχνολογίας ε, ως αυτοσκοπό, σκοπό. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και το να πούμε ότι η εκπαίδευση μπορεί να αντισταθεί θα σημαίνει ότι θα αγνοήσουμε τις εξελίξεις. Το να αγκαλιάσουμε λοιπόν την καινοτομία σημαίνει το να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους εκμάθησης, διδασκαλίας. Βέβαια η τεχνολογία δεν θα την τους δασκάλους γλωσσών και δεν θα μετατρέψει τους κακούς δάσκαλους σε καλούς. Ούτε πρόκειται για ένα μαγικό ραβδί που θα μετατρέψει τους μη ενδιαφερόμενους ή τους απρόθυμους μαθητές σε γρήγορους ε, ε, μαθητές ε, στις γλώσσες ή σε καλούς μαθητές. Ούτε καν η τεχνολογία θα μετατρέψει σε καλό διερμηνέα ένα φοιτητή ο οποίος δεν έχει το ταλέντο για τις γλώσσες και που δεν έχει την περιέργεια και γενικές γνώσεις. Όμως η τεχνολογία ήδη προσφέρει στους ε, εκπαιδευμένους δασκάλους και στους, ε, σε όσους έχουν όρεξη για μάθηση ένα πολύ πιο διευρυμένο περιβάλλον για μάθηση από η παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Είμαι βέβαιη πως η διδασκαλία των ε, διερμηνέων ε, σύντομα δεν θα είναι πια δυνατή χωρίς μια οθόνη. Δεν θα χρειάζεται σε λίγο καν να τους δείξουμε πώς θα συμβουλευθούν την ορολογία τους ε, online. Θα είναι ασύλληπτο το να τους προετοιμάζουμε στο μέλλον για συνεδριάσεις χωρίς έγγραφα. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε την τεχνολογία και την κοινοτομία με ανοιχτό μυαλό και να θα εκμεταλλευτούμε στο όσο μπορούμε περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του γοητευτικού κόσμου τη ε, διερμηνία συνεδρίων. Μπορώ λοιπόν μόνο να συγχαρώ τι ε, υπηρεσίε διερμηνία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων γιατί βρίσκονται στο ε, στην πρωτοπορία όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών στην ε, διοίκηση, στην κατάρτιση των διερμηνέων και στην επαγγελματική ζωή των διερμηνέων, με ικανοποίηση ε, διαπιστώνω πως οι υπηρεσίες μας σταθερά είναι τοποθετημένες ε, στην ε, πρωτοπορία, πρωτοπορία και ότι είναι έτοιμες πάντοτε να, να, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται. Αυτή η δραστήρια προσέγγιση είναι πολύ βασική ώστε να εξασφαλίσουμε πως η επόμενη γενεά διερμηνέων θα φτάσουν στην ε, απαιτητική αυτή αγορά πλήρως προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Σας εύχομαι κυρίες και κύριοι επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ αγαπητή Ανδρούλα για τα λόγια σας που πάντα είναι πηγή έμπνευση για όλους μας. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον Κλάους Βέλο, τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης έναν άνθρωπο που έχει πολύ πλούσια επαγγελματική σταδιοδρομία και πλούσιο βιογραφικό. Πέρασε από διάφορες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έφτασε στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχοντας γνώσεις για τη λειτουργία των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών και ξέρει εκ των έσω πολύ καλά τη λειτουργία του θεσμικού μας οργάνου. Ευχαριστώ θερμά και σου δίνω το λόγο, Κλάους. Ευχαριστώ πολύ κύριε <clears throat> Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε στα αγγλικά ο κύριος Σήμερα είναι μοναδική ευκαιρία που μας δίδετε και όχι μόνο μοναδική ευκαιρία για σας, αλλά και για μας. Για ποιο λόγο είναι μοναδική αυτή η ευκαιρία, γιατί μεταξύ ε, σας έχουμε 30 Πριτάνης που αυτό τον καιρό εκπαιδεύουν τους διερμηνείς του μέλλοντος. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ε, διερμηνείς όλο και περισσότερο είναι ένα αγαθό και βρισκόμαστε σε ένα ανταγωνισμό για τους καλύτερους ε, διερμηνείς σε πολλές γλώσσες και ακόμα περισσότερο αυτό θα ενταθεί μετά από 10 χρόνια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω μερικά επιχειρήματα γιατί ε, θα πρέπει να στείλετε τους καλύτερους φοιτητές σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω δέκα επιχειρήματα σας δώσω, ένα δεκάλογο. Πρώτο, βεβαίως, ε, ακαταμάχητο ήδη. Διότι ποιος δεν θα ήθελε να εργάζεται για ένα κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό βεβαίως, το επιχείρημα το μοιραζόμαστε με όλα τα θεσμικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Δεύτερο επιχείρημα. Με την Ευρώπη έχουμε το τελευταίο μεγάλο όραμα, το τελευταίο μεγάλο πολιτικό όραμα εν ζωή. Διότι μεγάλα οράματα είχαμε τον 20ο αιώνα, αλλά αυτά τα μεγάλα οράματα ήταν ολοκληρωτικά και γι' αυτό το λόγο απέτυχαν και έχουν ε, επιφέρει πολλά αρνητικά σε όλους μας. Το ευρωπαϊκό όραμα επέζησε διότι ακριβώ δεν είναι ολοκληρωτικό. Είναι ένα όραμα συνεργασίας, συμβιβασμού, συνύπαρξης και διαπραγματεύσεων. Τρίτο επιχείρημα. Βεβαίω όλα αυτά θα πρέπει να τα διαβιβάσετε στους φοιτητέ σας. Επιχείρημα τρίτο. Όποιος εργάζεται εδώ, εργάζεται στον τόπο που σήμερα συμβαίνουν οι αλλαγές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζουν τα πράγματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου. Μπορώ να σας παραθέσω λίγες μόνο από τις πιο πρόσφατες εμπειρίες μας. Έγινε τεράστια συζήτηση, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων στην Ευρώπη, για τις προτάσεις άκτα. Και πολλοί ε, συμμετείχαν ε, και πολιτικά και στο διαδίκτυο. Ποιος είχε το τελευταίο λόγο για την άκτα και αποφάσισε να μην προχωρήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις, οι μείζονες αποφάσεις. Σας ανέφερα μία που θα μπορούσα να προχωρήσω στο δημοσιονομικό κανονισμό. Εδώ είναι ο πιο ενδιαφέρον τόπος εργασίας, εάν σας ενδιαφέρει η πολιτική. Και επίσης, εδώ οικοδομούμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Όποιο ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση δεν μπορεί να βρει καλύτερο χώρο εργασία. 60 χρόνια αυτό κάνουμε. Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μα. Τώρα είμαστε συνομοθέτε επίση όρει και επίση ε, θα βεβαιωθούμε ότι θα ασκούμε το σωστό κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία όταν ε, πρόκειται για τις πολύ σημαντικές οικονομικές αποφάσεις και όλες τις αλλαγές που γνωρίζετε στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το τέταρτο επιχείρημα. Πέμπτον, εδώ στο κοινοβούλιο τα επιχειρήματα μετράνε. Δεν έχουμε σταθερή πλειοψηφία, ούτε σταθερή μειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε μια κατάσταση που ακριβώ επειδή κάποιο είναι στην πλειοψηφία έχει και δίκιο ή επειδή είναι στη μειοψηφία έχει άδικο από χέρι. Κάθε φορά, για κάθε νομοθέτημα, η πλειοψηφία χρειάζεται να σχηματιστεί βάσει επιχειρημάτων. Επιχείρημα έκτον. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, βλέπετε ε, επίπεδες ιεραρχίες. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι μας στη διοίκηση είμαστε πολύ πεπισμένοι για τη σημασία μας και όποιος έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, τον ε, επαναφέρει στην τάξη ένας ευρωβουλευτής πάρα πολύ γρήγορα. Έβδομο επιχείρημα. Μπορεί κανείς εδώ να ασκήσει επιχειρηματικό πνεύμα και θα πρέπει ε, να βασιζόμαστε σε αυτό. Αυτό κάναμε τα τελευταία 60 χρόνια, γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγα επίσημα δικαιώματα. Δηλαδή, η βασική ιδέα του Κοινοβουλίου ήταν ότι ε, δεν έχουμε καμία ευκαιρία, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Και βλέπετε ότι μετά από 60 χρόνια έχουμε προχωρήσει αρκετά επιχείρημα 8. Παρακαλώ να το διαβιβάσετε. Εδώ είναι θαυμάσιος χώρος για πολυεθνική και πολυπολιτισμική μάθηση. Δεν μην πάτε απλώς σε ένα συνέδριο για να συναντήσετε συναδέλφους σας από άλλες χώρες, αλλά καθημερινά εργάζεστε σε ένα περιβάλλον πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό από 27 κράτη-μέλη, 23 γλώσσες και ακόμα παραπέρα. Επιχείρημα ένατο εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να έχετε επαφέ με οποιαδήποτε γωνιά της γης. Το Κοινοβούλιο έχει αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο και επαφές και γνώσεις για όλο τον κόσμο και βεβαίως οι διερμηνείς συμμετέχουν πάρα πολύ ε, σε αυτή την προσπάθεια. Δέκατο και τελευταίο επιχείρημα και ελπίζω να σας πείσω και να μας στείλετε τους πιο καλούς σας φοιτητές ως Επαγγελματίε διερμηνέα. Γνωρίζετε κανένα άλλο μέρο στον κόσμο όπου θα πρέπει πάντα κανεί να εργάζεται σε ένα περιβάλλον 23 γλωσσών. Πουθενά. Δεν υπάρχει άλλο τόπο του κόσμου όπου να εργάζεται κανείς ε, διαρκώ και συστηματικά και ταυτόχρονα σε 23 γλώσσε. Αν ψάχνετε λοιπόν ε, ε, πιο συναρπαστική μορφή διερμηνίας πηγαίνετε και ελάτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Queridas, queridas amigas. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αφού ακούσαμε την Επίτροπο Βασιλείου και τον κύριο Βέλε, τον Γενικό Γραμματέα, που δεν ξέρω ίσως πρέπει να φύγουν ε, και ίσως φύγουν στη διάρκεια της δικής μου ομιλίας, γιατί τώρα θα σας παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις ως πολιτικός ηθήνων. χωρίς δηλαδή τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς ε, που αντιμετωπίζουν άλλες κατηγορίες. Ε, η διοίκηση, για παράδειγμα, δεσμεύεται από μια υποχρέωση διπλωματικής έκφρασης. Εγώ δεν υπόκειμαι σε τέτοιο περιορισμό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, εκφράσω την, το θαυμασμό μου για αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι και ε, δεν θα επαναληφθεί και όλα, αλλά με ανθρώπους σαν την Όλια Κοσμίδου ακόμη και τα θαύματα επαναλαμβάνονται. Αλλά πραγματικά τέτοιου είδου ε, οργάνωση δεν είχα ξαναδεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι χρόνια ολόκληρα Ευρωβουλευτή. και ιδιαίτερα με τέτοιο αντικείμενο. Είναι πραγματικά εξαιρετική ευκαιρία, καταπληκτική, για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και να παρουσιάσουμε και κάποιες σκέψεις και αυτή την ευκαιρία θα την ε, αδράξω και εγώ τώρα. Καταρχήν, θεωρώ ότι η πολυγλωσία και ήταν ανέκαθεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα εξαιρετικά σημαντικό φαινόμενο, ένα ζωτική σημασία φαινόμενο και ένα, μια ένδειξη ε, δημοκρατικής ταυτότητας. Αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι χάρη στην δημοκρατική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφυσούμε δημοκρατία και στα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα που είτε επειδή είναι δημοκρατικά, επειδή έχουν άλλη φύση, δεν έχουν ούτε τα χαρακτηριστικά αυτά, ούτε την ανάγκη αυτή. Θα ήθελα επίσης να σας εξηγήσω πώς βιώνουμε στην πράξη την πολυγλωσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας εκθέσω και κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Επίσης θα σας παρουσιάσω τρόπους υπερκέρασης αυτών των δυσκολιών. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ε, στην προσπάθειά μου να εξηγήσω μερικές δυσκολίες, ίσως το κάνω κάπως ε, απότομα και ομά, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να σας κατακτήσουμε, γιατί είστε οι απαραίτητοι μας σύμμαχοι στο καθήκον που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο δικό μου καθήκον, δηλαδή να λειτουργήσει πραγματικά ε, υποκαθεστώς πολυγλωσία στο θεσμικό μας όργανο. Θα σας εξηγήσω καταρχήν πώς λειτουργούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αναφυσβήτητα το μοναδικό θεσμικό όργανο στο παγκόσμιο προσκήνιο που χρησιμοποιεί τόσο πολλές γλώσσες. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το όργανο που χρησιμοποιεί τις περισσότερες γλώσσες. Στο περίπλοκο αυτό ευρωπαϊκό πλέγμα και διάρθρωση δεν έχουμε άλλο θεσμικό όργανο που να λειτουργεί με βάση αυτή τη μέρημνα και την επιτακτική ανάγκη της λειτουργίας υπό πολυγλωσσικό καθεστώς. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε γλώσσες εργασίας. Κάτι που άλλα θεσμικά όργανα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν. Και είναι λογικό. Το αν είναι λογικό να τις έχουν ή όχι είναι άλλο θέμα δεν πρόκειται να επισέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς πάντως, όταν λέω ότι δεν έχουμε γλώσσες εργασίας, ίσως κάνω λάθος, γιατί έχουμε 24 γλώσσες εργασίας. Δεν είναι 23 οι γλώσσες εργασίας μας, είναι 23, αλλά ήδη χρησιμοποιούμε και τα κροατικά. Γιατί ήδη προεξοφλούμε την κατάσταση που θα δημιουργηθεί μετά από λίγους μήνες. Γιατί αν δεν χρησιμοποιούσαμε ήδη τα κροατικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν θα μπορούσαμε ε, τη στιγμή της ένταξης Κροατίας σε λίγους μήνες να μετατραπούν ε, νύχθη μερό και τα κροατικά σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και κάνουμε τη σχετική προεργασία. Εργαζόμαστε λοιπόν με 24 γλώσσες, αλλά όχι μόνο με 24 γλώσσες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βλέψεις να μετατραπεί σε πολύ σημαντικό ε, παράγοντα διεθνώς. Και ως τέτοιος ε, διεθνής παράγοντας, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεργασία με άλλους ε, διεθνεί παράγοντε με εταίρους, με συνεργάτες σε αυτό το καθεστώς της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γι' αυτό και σχεδόν μονίμως χρησιμοποιούμε και τα ρωσικά και τα αραβικά και τα κινέζικα και μερικές φορές και άλλες γλώσσες ανάλογα με τις συναντήσεις που έχουμε, με τις συνεδριάσεις που έχουμε, γιατί ε, φιλοξενούμε και ε, εκπροσώπους ε, άλλων χωρών ή μετέχουμε στις συνεδριάσεις με ηθήνοντες και άλλων χωρών και έτσι χρησιμοποιούμε και άλλες γλώσσες. Κάτι που ισχύει άλλωστε και στη σημερινή εκδήλωση. 24 αυτές λοιπόν γλώσσες, τις οποίες λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις οποίες χρησιμοποιεί ως γλώσσες εργασίας, προϋποθέτουν μια τεράστια προσπάθεια όχι μόνο για τη λειτουργία τους, όχι μόνο δηλαδή τη λογιστική προσπάθεια, τη μηχανική. <laughs> Μερικές φορές μιλάμε ε, για τα ενιδρία που μοιάζουν οι καμπίνες και πραγματικά έχουμε και το πιο σημαντικό ενιδρίο, το πιο σημαντική καμπίνα που είναι των τεχνικών και που εξασφαλίζει τι ε, συνδέσει. Είναι σημαντική ε, λοιπόν οι καμπίνε διερμηνία, τα ενιδρία τη διερμηνία, αλλά πολύ σημαντικό είναι και το ενιδρίο των τεχνικών, που χάρη στη δική του συνεισφορά φτάνουν ε, οι καμπίνε από, τις, από του διάφορου τεχνικού διάβλου και μπορεί κανεί να ακούει τη γλώσσα του. Έχουμε και το θέμα της πρόσληψης φυσικά των, διερμηνέων, αλλά μην ξεχνούμε και τη μεγάλη σημασία που έχουν και οι μεταφραστές, γιατί είμαστε ένα θεσμικό όργανο στο οποίο κάθε λέξη που προφέρεται, κάθε λέξη που ακούγεται, γιατί σε ένα, ευρωπαϊκό, σε ένα κοινοβούλιο ακούγονται πολλές α, λέξεις, κάθε λέξη λοιπόν που προφέρεται και που ακούγεται ταυτόχρονα ε, ερμηνεύεται και μεταφρα, ε, ε, σε άλλες 23 γλώσσες. Και κάθε, ε, γλώσσα, κάθε λέξη που προφέρεται ταυτόχρονα επίσης ε, πρέπει να μεταφραστεί και στις υπόλοιπες γλώσσες. Από το πρωτότυπο στις υπόλοιπες. Κάτι τέτοιο δημιουργεί τεράστιες τεχνικές περιπλοκές και προϋποθέτει έναν τεράστιο επαγγελματισμό των αρμοδίων και αυτών που ε, κάνουν, εξασφαλίζουν τη διαχείριση αλλά και αυτών που υλοποιούν αυτό το έργο. Ο Κλάους Βέλε είπε ότι ε, που έχει, είναι πολύ διακριτικός άνθρωπος και έχει πάρα πολλά προσόντα. Δεν είπε ότι οι, οι διερμηνείς και οι μεταφραστές ανήκουν σε ένα επάγγελμα στο οποίο δεν υπάρχει ανεργία. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου στις περισσότερες χώρες η ανεργία είναι σημαντική μάστιγα. Σε αυτό το επάγγελμα του μεταφραστή και του διερμηνέα δεν υπάρχει ανεργία. Βέβαια, εντάξει, δεν έχουν ε, τα κασέ που έχουν ε, κάποιοι ποδοσφαιριστές ή αστέρια του πενταγράμμου. Αλλά πάντως σίγουρα έχουν πολύ καλές συνθήκε εργασίας και πιστεύω ότι πραγματικά το επάγγελμα του διερμηνέα και του μεταφραστή είναι ένα καταπληκτικό επάγγελμα και μάλιστα είχα το, την τιμή να το ασκήσω στην <laughs> προσωπική μου ζωή για χρόνια ολόκληρα και πιστεύω ότι είναι ένα καταπληκτικό επάγγελμα και νομίζω ότι μπορούμε να, να προσελκύσουμε νέους να διδαχθούν και να ασκήσουν μετά αυτό το επάγγελμα. Επίσης, το φαινόμενο της διερμηνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σχεδόν μαγικό φαινόμενο. Είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές, γιατί μου συμβαίνει σχεδόν καθημερινά. Εμείς, οι Ευρωβουλευτές, λαμβάνουμε ε, και υποδεχόμαστε σημαντικό ρυθμό επισκεπτών από τις πατρίδες μας που έρχονται για να δουν πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν έρχονται ένας-δύο, έρχονται 20-30% συμπατριώτες μου, άνδρες και γυναίκες κάποιου μέσου επίπεδου, που συνήθως μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Και είναι αυτό σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα θεσμικά όργανα, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχονται λοιπόν 30 συμπατριώτε μου. Κάθονται εδώ όπω καλή ώρα κάθεστε κι εσεί. Και του λέω, βάλτε τα ακουστικά, γυρίστε στο 8 και θα ακούσετε τη γλώσσα σα. Και ενώ είναι φυσιολογικά οι άνθρωποι κάτω, ξαφνικά είναι σαν να, σαν να παθαίνουν κάτι. Και μου λέει κάποιο, πώ είναι δυνατόν α, <laughs> αυτή, να, μην, να ακούμε να μιλάει μια κυρία και να ακούγεται μια αντρική φωνή Πώς είναι δυνατόν ε, να βλέπουμε να μιλεί άντρε και να ακούμε μία φωνή σοπράνο. Μα τους εξηγώ, δεν ακούτε τον ίδιο μιλητή. Μπορεί να είστε δυο εδώ, αλλά ποτέ δεν ακούσετε απευθεία τον ομιλητή. Ακούσατε, βλέπετε στην καμπίνα 8, εκεί που έχει τον αριθμό 8. Εκεί είναι η ισπανική καμπίνα. Ακούσατε εκείνο τον κύριο και εκείνη την κυρία που βρίσκονται στην καμπίνα και που εναλλάσσονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχεδόν ε, μία μαγική ικανότητα, ένα καταπληκτικό ταλέντο να ακούν μία γλώσσα στα αυτιά τους και να την μετατρέπουν στην μητρική τους γλώσσα, στη γλώσσα που εσείς ακούτε. Οπότε οι άνθρωποι πραγματικά μένουν εμβρόντιτοι. Μένουν εμβρόντιτοι γιατί καταλαβαίνω ότι χάρη σε αυτό το μηχανισμό είναι πραγματικά πολίτες και νιώθουν πολίτες. Σε ελάχιστες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι άνδρε και οι γυναίκε που εκεί διαβίουν ανέκαθεν αισθάνονται ότι ήταν πολίτε. Εμεί δεν είχαμε πάντα αυτή την εμπειρία. Μερικέ φορέ ε, δώσαμε τη ζωή μα και το αίμα μα για να αποκτήσουμε αυτή την ιδιότητα του πολίτη. Χρειάστηκε να δώσουμε τη ζωή μα, να θυσιάσουμε τη ζωή μα για να διεκδικήσουμε την ιδιότητα του πολίτη. Να έχουμε το δικαίωμα δηλαδή, να έχουμε γνώμη για τη μοίρα μα, για το πεπρωμένο μα και να μπορούμε να ελέγχουμε του ηθήνοντέ μα, ε, αυτού που εκλέγουμε για να προασπίσουν τα συμφέροντά μα. Αυτό συμβαίνει όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οποιοδήποτε Ισπανός, οποιοδήποτε συμπατριώτης μου μπορεί να έρθει και να ακούσει τι συζητάτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούει εμένα που μιλάω τα Ισπανικά, αλλά ακούει και τους υπόλοιπους και μπορεί να τους ακούσει και εκείνους στα Ισπανικά. Και είναι ένα θέμα που το αναφέρω συχνά σε ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζουν σε ένα πολύ κλειστό κόσμο που όλοι μιλάνε αγγλικά. Δεν ξέρω κανέναν υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μην μιλάει αγγλικά. Ούτε έναν. Και φυσικά, όταν κανεί ζει στον κόσμο του, όπου όλοι μιλάνε σε μια ε, φούσκα που όλοι μιλάνε ε, αγγλικά, μπορεί να πιστεύουν μετά από λίγο καιρό ότι όλο ο κόσμο μιλάει αγγλικά. Και πραγματικά δεν ισχύει αυτό. Ούτε στον κόσμο, ούτε καν μέσα στην Ευρώπη. Στην πατρίδα μου την Ισπανία μόνο το 5% των Ισπανών μιλάνε άψογα αγγλικά ή πολύ σωστά τα αγγλικά και 15% επιπλέον καταλαβαίνουν κουτσά στραβά τα αγγλικά. Δηλαδή 80% των Ισπανών πολιτών δεν έχει καμία γνώση, είναι τελείως ανίκανο να παρακολουθήσει τις συζητήσεις που γίνονται στα αγγλικά και δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν γινόταν μόνο στα αγγλικά. Αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι συζητήσεις γίνονται με τρόπο που γίνεται προσιτός και για τους πολίτες. Πραγματικά λοιπόν ζούμε σε ένα θεσμικό όργανο που είναι αμυγός δημοκρατικό. Γιατί αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε να ακούουν οι συμπολίτε μας να παρακολουθούν και να ελέγχουν αυτό που συμβαίνει, τότε πώς θα εστερνιστούν αυτό το σχέδιο, πώς θα το οικειοποιηθούν, πώς θα καταλάβουν ότι αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν είναι σχέδιο γραφειοκρατών και ευρωβουλευτών, αλλά να το νιώσουν δικό τους. Για να το κάνουν κτήμα τους, οι συμπολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν βήμα προ βήμα αυτό που συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα στη μόνη γλώσσα που του είναι προσιτή, που είναι η μητρική του γλώσσα. Και αυτό σα το λέω για την Ισπανία, αλλά δεν είναι ε, κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ισπανία, συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. Μπορεί σε τρει-τέσσερι μόνο χώρε που ε, αντί να μιλάμε για 20-25% ε, που μιλάνε αγγλικά, να μιλάμε για 30%. Μόλις επέστρεψα από την Κύπρο. Εκεί πραγματικά για, πολύ για πολλά χρόνια πιο πιοκρατικό καθεστώ και πολλοί μιλάνε αγγλικά. Αλλά από του τρει ε, ε από τον Πατριάρχη, ε, τον Αρχιεπίσκοπο, κανένα δεν μιλούσε αγγλικά ή τουλάχιστον με πολλέ δυσκολίε. Δεν είναι ότι μιλάνε όλοι, ούτε καν στην Κύπρο αγγλικά. Μου έλεγαν are there, better, half, half an hour. Ε, ε δεν μπορεί κάποιο με τόσο στοιχειώδη αγγλικά να παρακολουθήσει τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να σα πω, εν πάση περιπτώσει, από την αρχή. Πώ λειτουργούμε και γιατί. Εδώ και λίγη ώρα σα μιλάω και για τις δυσκολίες, γιατί έχουμε κάποιες δυσκολίες και κάποιες αντιστάσεις, μερικές φορές ακόμη και κάποια εχθρότητα. Για παράδειγμα, ο κόσμος μας λέει ότι στοιχίζει πολύ ακριβά η διερμηνία και η μετάφραση. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι δαπανηρή και η μετάφραση και η διερμηνία. Αλλά η διερμηνία και η μετάφραση κοστίζουν πολύ λιγότερο από ότι τα μέσα μαζικής, μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εχθρικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σκανδαλοθυρικά και κάνουν καταγγελίες, ισχυρίζονται ότι είναι πολύ ακριβή η μετάφραση και η διερμηνία Στοιχίζουν όμως αυτό που θα στοίχιζε ένα καφέ το χρόνο ένα Ευρωπαίο πολίτη. Μπορεί να είναι κάποιο ποσό, αλλά δεν είναι και κανένα υπέρογκο ποσό. Πολλό δε μάλλον που έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε 500 εκατομμύρια πολίτες. Γιατί σε ποια χώρα μπορεί κανείς να πιει καφέ με ένα ευρώ. Στην Ισπανία δεν είναι πια εύκολο κάτι τέτοιο. Εδώ το πληρώνουμε 70 ε, λεπτά γιατί επιχορηγείται. Αλλά πραγματικά τόσο είναι το κόστος ε, της μετάφρασης και διερμηνίας. 500 εκατομμύρια σε, όλες τις, ε, όλα τα επίπεδα και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό, είναι ένα είδος φόρου της δημοκρατίας που είναι ανεκτήμητη, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήματα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι απαραίτητη η διερμηνία, είναι πολυτέλεια, είναι ιδιοτροπία, είναι ένα καπρίτσιο. Σας είπα όμως ότι είναι απαραίτητη για να κρατήσουμε την, την, την ταυτότητά μα και να μπορέσουν οι πολίτες να εστερνιστούν να κάνουν κτήμα στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Και λένε ότι μερικές φορές δεν χρειάζονται διερμηνεί και μεταφραστέ γιατί μπορεί η μετάφραση να γίνεται μηχανικά, με μηχανέ. Εντάξει, γράψτε μου σε μισή σελίδα μερικές φράσεις. Να, το, να τις βάλουμε στο Google Translation, στη μετάφραση του Google. Να σας βγει αυτόματη μετάφραση μηχανική και να μου πείτε αν καταλαβαίνετε έστω και λέξη από αυτά που διαβάζετε. Δεν ξέρω σε 30 χρόνια τι ικανότητα θα έχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί όντως, ε, πριν από 30 χρόνια σημερινές εξελίξεις ήταν αδιανόητες. Πάντως σήμερα Ούτε η δερμήνια, ούτε η μετάφραση μπορεί να γίνει μηχανικά και αυτόματα. Παρόλο που έχουμε εξέλιξη ραγδαία των νέων τεχνολογιών και πολύ εύστοχα και πολύ γλαφυρά και παραστατικά μας μίλησε η Επίτροπος για τις νέες τεχνολογίες και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ανάγκη χρησιμοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες και είμαστε και πρωτοπόροι στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Μάλιστα προσφέρουμε ε, και στις υπηρεσίες μας, ε, τις υπηρεσίες μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ομένα Έθνη που ζητούν την υπηρεσία μας και έχουμε και γραπτές συμβάσεις με άλλα όργανα. Γιατί από την εμπειρία μας ε, που δουλεύουμε με 23, 24, 25, 27 γλώσσες έχουμε τεράστια πλούσια εμπειρία και γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και τα νέα μηχανήματα και τις νέες τεχνολογίες. Και έχουμε και συνεχή σχέση και επαφή με τη βιομηχανία, με τον κλάδο. Γιατί ο κλάδος από μόνος του ουδέποτε δεν θα φανταζόταν ότι θα υπήρχε ένα όργανο που θα χρειαζόταν επικοινωνία σε 25-26 και γλώσσες. Αυτή η επικοινωνία λοιπόν διασφαλίζεται συνεχώς με τους αρμοδίους του κλάδου και έχουμε εμπειρογνώμονες που έρχονται εδώ και κάνουν ε, ασκήσεις, κάνουν στάζ, παρακολουθούν σεμινάρια, βλέπουν πού μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες καμπίνες. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο αριθμός των ενηδρίων είναι πεπερασμένος. Δεν θα έχουμε χρόνο να προσθέσουμε νέες καμπίνες. Βέβαια, μερικές φορές δεν συμφωνούν μαζί μου οι διερμηνήσεις. Χρειαστεί να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να μην, μείνουν, ε, να μην είναι στην ίδια αίθουσα. Καλό είναι να μας βλέπουν, αλλά ίσως κάποια στιγμή δεν θα είναι μέσα στην αίθουσα, αλλά θα είναι κάπου κοντά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν Όσο είχα να σας πω προς το παρόν. Πάντως, η προάσπιση της πολυγλωσσίας ε, περνάει φυσικά από την προαγωγή της διερμηνίας και της ε, μετάφρασης, αλλά και την προαγωγή της μελέτης, ε, της διδασκαλίας και της εκμάθησης των γλωσσών και την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών. Ευτυχώ η, κυρία Επίτροπος έχει συμπεριλάβει αυτά τα θέματα σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι μια ευαισθητοποίηση που θα πρέπει να γίνει, μια συνειδητοποίηση. Γιατί για πολλά χρόνια ακόμη δεν θα έχουμε πάνω από 20-25% των Ευρωπαίων πολιτών που θα είναι ικανό να παρακολουθεί τι κάνουμε σε όλες αυτές τις γλώσσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, αν δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στη γλώσσα του. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάποιες τολμηρές σκέψεις, γιατί ε, έκανα κάποιες σκέψεις για το τι περνάει αυτόν τον καιρό η Ήπειρός μας. Και δεν σας μιλώ εδώ σε αρμόδιες πολλές γνωσίες, αλλά σας μιλώ για το ίδιο το ευρωπαϊκό όραμα, το ευρωπαϊκό σχέδιο, γιατί είμαι από τους αντιπροέδρους που έχουν αυτή την αρμοδιότητα να προωθήσει αυτό το σχέδιο, ξεπερνώντας τις δυσκολίες. Το σχέδιο λοιπόν της ευρωπαϊκής οικοδόμησης διανύει μια δύσκολη στιγμή, περίπλοκη. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης φυσικά είναι πολύ σημαντικό και θα είναι πραγματικά ε, θα μας δώσει μια σημαντική όθηση για να κρατήσουμε την πορεία μας. Θα είναι σημαντικό εφαλτήριο και εντάξει την πορεία την έχουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε κάπως ε, την πορεία μας. Βέβαια ο ρυθμός μπορεί να σταματήσει και η κατεύθυνση να στραβώσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσουμε και την κατεύθυνση ε, σταθερή και το ρυθμό μας αμύωτο. Αλλά πραγματικά διανύουμε μια κρίση πολύ ε, σκληρή που δεν είναι μόνο οικονομική και χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική. Είναι μια κρίση που ε, κάνει ώστε αυτό το σχέδιο που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια και συνεχίζει να επιβιώνει ως αλληλέγγυο σχέδιο, αρχίζει και μετατρέπεται δυστυχώ σε ένα σχέδιο που δεν χαρακτηρίζεται πια από αλληλεγγύη. Το σχέδιο αυτό ήταν αρχικά ένα σχέδιο αλληλεγγύης και πηγή έμπνευση ε, για τις χώρες και για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Αυτό το σχέδιο όμως που ήταν κατεξοχήν σχέδιο αλληλεγγύης δημιούργησε τεράστια συμπάθεια, ενθουσιασμό και προσδοκίες σε πολλές χώρες που χάρη σε αυτή την αλληλεγγύη κατάφεραν να αναβαθμίσουν το βιωτικό τους επίπεδο και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Στο μέτρο όμως που αυτό το αρχικά αλληλέγγυο σχέδιο θα μετατραπεί σε μία αλληλέγγυο σχέδιο, στο μέτρο που παρακολουθούμε μία έξαρση του εγωισμού και του εθνικισμού που θέτει σε κίνδυνο την ταυτότητα αυτού του αρχικά αλληλέγγυου σχεδίου, αυτό που παρατηρούμε είναι μία πολύ επικίνδυνη ε, και ε, έντονη απόρριψη των Ευρωπαίων πολιτών κατά το σχέδιο αυτού, στο μέτρο που αυτό γίνεται αναλληλέγγυο. Πριν από τρεις μέρες ε, ήμουν στο Johannesburg και το λέω πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση και ανατριχιάζω. Ήμουν στην συνεδρίαση που έχουμε κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Παναφρικανική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται τα κοινοβούλια όλων των χωρών της Αφρικής με ε, ανθρώπους με όλο και πιο μεγαλύτερες ελευθερίες, δεξιότητες ε, και πιο εκλεπτισμένους. Τους μιλούσε λοιπόν για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Φαντάζομαι πολύ είναι εξοικειωμένοι με το θέμα αυτό και κάποια στιγμή μου έδωσαν ένα χαρτί, ήμουν στο βήμα και μου δίνουν ένα χαρτί που ε, έλεγε την πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Διέκοψα τότε την ομιλία μου και είπε μόλις έμαθα, κυρίες και κύριοι, αυτό και αυτό. Και η αίθουσα που ήταν μεγαλύτερη από εδώ, ε, όλοι σηκώθηκαν αυτόματα όρθιοι και για τέσσερα λεπτά χειροκροτούσαν. Νόμιζα πραγματικά ότι θα καταρρεύσω μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν το άντεξα. Για τέσσερα λεπτά όρθιοι Αφρικανοί χειροκροτούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά το 80% οι άνθρωποι αυτοί ε, έδωσαν μάχη και πλήρωσαν πολύ ακριβά τον αγώνα τους, όχι μόνο εξαιτία τη σκλάβια, τη της ε, αλλά και εξαιτία των απεικιοκρατικών βλέψεων της Γαλλίας, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και ξαφνικά ακριβώς αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκατέστησε την ειρήνη σε μια ήπειρο που είχε καταρακωθεί από τον όλεθρο του πολέμου και ξεχνώντας αυτή την ζωφερή απεικιοκρατική περίοδο και παρελθόν, αυτοί οι άνθρωποι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν. Εμείς θα δημιουργήσουμε και το Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αλλά είδα ότι αυτοί οι Αφρικανοί αναγνώρισαν ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχέση με την παλιά απεικιοκρατική Ευρώπη. Είναι μια δύναμη που είναι πηγή έμπνευση για αυτούς, για την ε, συνεργασία τους, για το τέλος των πολέμων, για την ευημερία, για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιος Ευρωπαίος δεν θα ανατριχιάσει και δεν θα συγκινηθεί βαθύτατα με αυτά που λέω. Πραγματικά, αν μένει ασυγκίνητος, δεν αξίζει να λέγεται Ευρωπαίος. Σε καμία περίπτωση δεν θα έμενα συγκίνητος ο Ευρωπαίος ή η Ευρωπαία του σήμερα αλλά και του αύριο. Πραγματικά συγκινούμε και τώρα που το ξαναθυμάμαι, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι κανείς και όσο πιο ε, μεγάλος γνώση για την ιστορία, μένει και πιο εύκολα, συγκινείται και πιο εύκολα από τέτοιε εκδηλώσεις. Όλα αυτά λοιπόν με συγκινούν, με εμπνέουν σε αυτό το περιβάλλον της πολυγλωσσίας που πραγματικά είναι σημαντική όθηση για την δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την συνεργασία των λαών και για το μεγαλύτερο ανθρωπισμό. Θα ήθελα να σας, ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπομονή σας και για την προσοχή με την οποία παρακολουθήσατε την ομίλια μου. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Θα χαιρετήσουμε την κυρία Βασιλείου και τον κύριο Βέλε. Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Δεν ξέρω πώς θέλετε τώρα αμέσω να ε, πούμε στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα, στο πρώτο κεφάλαιο της διάσκεψης μετά την εναρκτήρια αυτή ενότητα.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 Σύντομα, μια πρακτική σημείωση. Έχετε όλοι στα έδρανά σας μια σημείωση για τη διερμηνία. Βλέπετε ποιες γλώσσες ακούτε, μπορείτε να ακούτε και τις ε, καμπίνες και εκτός αυτών αραβικά, κινέζικα και τουρκικά. Μπορείτε να μιλήσετε, όχι να ακούσετε. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενη ενότητα της σημερινής διάσκεψης και με μεγάλη χαρά έχω την ευκαιρία να καλωσορίσω το διευθυντή του Euronews, τον κύριο Φιλίπ Κέιλα, ο οποίος θα αναλάβει αυτή τη στιγμή την ε, υπόθεση του συντονισμού της συζήτησης. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και την κυρία Κοσμίδου για την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε η Euronews είναι ε, ο τηλεοπτικός σταθμός της πολυγλωσσίας και αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα εδώ σας στο σπίτι μας. Βέβαια εμείς ένα μέσο ενημέρωση είμαστε, δεν είμαστε πανεπιστήμιο, αλλά έχουμε 400 δημοσιογράφους που μοιρούν 23 γλώσσες και ε, εκφράζονται σε 11 γλώσσες σε όλο τον κόσμο και συνηθίζουν να συζητούν για θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μεταδίδουν και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε ένα ε, πολύ ε, γλώσσο πλαίσιο. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα πήγα στην Ινδία και διαπίστωσα και το Ινδικό Κοινοβούλιο είναι πολύγλωσσο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντίστοιχα πολλά τέτοια κοινοβούλια, αλλά και στην ε, ε, Ινδική Βουλή έχετε ε, επίσημες γλώσσες και 20 μάλιστα επίσημες γλώσσες. Δεν μιλούν όλοι στην Ινδία αγγλικά, ούτε Ινδί. Υπάρχουν και άλλες γλώσσες από το Κασμίρ και όπως οι ευρωβουλευτές και οι Ινδοί βουλευτές εργάζονται με ακουστικά και με διερμηνείς. Και η πολυγλωσία είναι ίσως πιο διαδεδομένη από ό,τι ε, φαίνεται εκ πρώτης όψης. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Στεφάν Λόπες που ε, είναι μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διεθνή Οργανισμό της ε, Φραγκοφωνή, της Γαλλομάθειας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ε, θαυμάσιας αυτής εκδήλωσης. Όπως είπε προηγουμένως ο βουλευτής κύριος Μαρτίνες, είναι υπέροχη αυτή η ευκαιρία που έχουμε σήμερα. Εσείς είστε όλοι εκπρόσωποι ε, της ε, εκπαίδευσης, είμαστε στο κοινοβούλιο που είναι ε, αυτός ο ναός της δημοκρατίας και ταυτόχρονα ε, μαζί με εσά, κυρίες και κύριοι Πριτάνη συζητούμε το μέλλον και με μεγάλη χαρά παίρνω το λόγο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα να παίρνει κανείς το λόγο μετά από αυτόν τον ρήτορα, τον Ευρωβουλευτή κύριο Μαρτίνες με την τόσο εμπνευσμένη ομιλία του και με τόσο πάθος. Θα ήθελα εγώ λίγο να σας μιλήσω για την ε, πολυγλωσία στο κοινοβούλιο, την ποικιλομορφία, τη διάβρωσή της, αλλά ε, και τέλος να δούμε και τι διακυβεύεται και πώς μπορεί να διαφυλαχθεί και να ε, διασωθεί στις κοινωνίες μας η πολυγλωσία. Οι κοινωνιογλωσσολόγοι αξιολογούν την διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία των γλωσσών στον κόσμο σε 7.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις πανεπιστημιακές σχολές. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην κατανομή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υπήρους. Υπολογίζεται περίπου 32% ε, είναι γλώσσες ε, της Ασίας, 30% στην Αφρική, 19% στο χώρο του Ειρηνικού ωκεανού γιατί δεν είναι Ήπειρος, 15% στην Αμερικανική Ήπειρο και στην Ευρώπη που βρισκόμαστε στην καρδιά της πολυγλωσσίας αυτό ε, αντιπροσωπεύει μόλις το 3%. Δηλαδή ε, πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί απέναντι σε εκπροσώπου άλλων υπήρων που έχουμε ορισμένου ε, εδώ ενώπιον μας. Αυτό που μας προβληματίζει αρκετά είναι το εξή. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μια ήπειρο και όσο πιο περισσότερο καιρό είναι ανεπτυγμένη, τόσο λιγότερες γλώσσες ομιλούνται στην ήπειρο αυτή και αυτό είναι παράδοξο. Έτσι, εκ πρώτης λίγο ενισχυτικό και μας προβληματίζει. Ε, ορισμένοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στη βιοπικιλότητα και τη γλωσσική ποικιλότητα. Σε υπήρους και σε περιοχές όπου η βιοπικιλότητα απειλείται, υποχωρεί και η ίδια η γλωσσική ποικιλότητα και είναι πιο αδύναμη. Και αυτό πραγματικά μας προβληματίζει και μας ανησυχεί από πολλές πλευρές. από τις 7.000 γλώσσες, οι 4.800 διατηρούνται σε περιοχές που είναι πλούσιες σε βιοπικιλότητα. Άρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ βιοπικιλότητας και γλωσσικής ποικιλία. Μεταξύ αυτών λοιπόν των γλωσσών, 26,5% ομιλούνται ε, από κοινότητες 10.000 ε, έως 100.000 ατόμων, 29,4% από κοινότητες 10.000 έως 1.000 ατόμων και 27% από μικρές κοινότητες από 1.000 μέχρι 100 ομιλούντες τη γλώσσα αυτή κάθε φορά. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, για να μην πω στις τρεις, είναι προφανές ότι Πολλέ από αυτές τις γλώσσες, για να μην πω η μεγάλη του πλειονότητα, απειλούνται. πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα και σίγουρα μακροπρόθεσμα. Υπολογίζεται 50 με 90% των γλωσσών αυτών και εδώ κυμαίνονται οι εργασίες ανάλογα με το πανεπιστήμιο ενδεχομένως να εξαφανιστούν πριν το τέλος του 21ου αιώνα. Πέρα λοιπόν από ε, αυτές τις κινδυνολογίες, το θέμα είναι να καταλάβουμε πώς διαβρώνεται μία γλώσσα. Οι εθνολόγοι υπολογίζουν ότι αυτό συνδέεται με τους διάφορους τρόπους που προσλαμβάνει η πολιτική οργάνωση, η κοινωνική οργάνωση και η οικονομική οργάνωση του κόσμου. Από τι χαρακτηρίζεται αυτή από φαινόμενα εξορθολογισμού, συγκέντρωσης, τυποποίησης, δηλαδή δημιουργίας κανόνων και προτύπων και όλα αυτά οδηγούν ε, σε μια μορφή ε, πολιτικής συγκέντρωσης. Ε, κράτη, διακρατικές δομές, πολυμερείς, οικονομική παγκοσμιοποίηση αστική ανάπτυξη και αστιφιλία, ε, συγκέντρωση κοινωνική ε, σε πόλεις. Βέβαια, αυτή η διαδικασία που περιγράφω εδώ σε αυτό το ειρηνικό κοινοβούλιο και φιλικό δεν είναι πάντα ειρηνική και ούτε είναι άσχετη με συσχετισμού δυνάμεων. Και αυτό ο συσχετισμός δυνάμεων οδηγεί σε μια επιλογή που δεν είναι κατά ανάγκη φυσική επιλογή, είναι πολιτιστική επιλογή, η οποία ε, παράγει πολιτιστικό αποκλεισμό και τελικά περιορισμό και μείωση της διαφορετικότητας και της ποικιλία. Ένας αριθμό γλωσσών έτσι αποκλείονται από την δημόσια έκφραση μιας ανθρώπινης κοινότητας και είτε εξαφανίζονται είτε περιθωριοποιούνται. Οκτώ γλώσσες ομιλούνται σήμερα από ε, πολυάριθμες κοινότητες, πολυπληθείς, ε, που απαρτίζονται από εκατομμύρια και πλέον των ομιλούντων. Είναι τα κινέζικα, τα αγγλικά, μαλισιανά, ισπανικά, πορτογαλικά, αραβικά, γαλλικά και ίντι. Ορισμένες από τις γλώσσες αυτές ομιλούνται από τις κοινότητες σε πιο τοπικό επίπεδο είναι ε, εντός μίας ε, κρατικής οντότητας. Ενώ άλλες γλώσσες είναι πιο διαδεδομένες σε πολλά κράτη, σε πολλές υπήρους. Και οι γλώσσες αυτές, οκτώ που σας ανέφερα, ε, μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις ομάδες διάδοσης. Τα κινέζικα, τα μαλαισιανά και τα ίντι ανήκουν σε μια ομάδα που την ονομάζουμε σούπερ κεντρική αλλά εντοπισμένη τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα αραβικά και τα γαλλικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αλλά είναι πιο διαδεδομένα γεωγραφικά για τους ε, απικιακούς λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Και τα αγγλικά, που έχει φτάσει σε ένα επίπεδο υπερκεντρικό, υπέρ σαντραλ, όχι σούπερ σαντραλ. Δηλαδή το ξέρουμε και όχι μόνο για λόγους απικιοκρατίας αλλά ε, από ό,τι φαίνεται τα αγγλικά πέρα από τη γλώσσα που ήταν και που συνέδε μια ε, πολιτιστική κοινότητα, η πολιτισμική, ε, έχει γίνει πλέον ένας κοινωνικός κώδικας που έχει επιβληθεί πλέον όχι μόνο σε μια σειρά από θεσμού και ο βουλευτής κύριος Μαρτίνε αναφέρθηκε σε αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο έχει επιβληθεί στα θεσμικά τη όργανα, αλλά δεν αφορά μόνο ε, την Ένωση και ισχύει και αλλού αυτό και στον ΟΗΕ, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας, εκτοπίζοντας ε, τις άλλες γλώσσες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η ε, φυσική διαδικασία ε, κοινωνικής ανέλυξης που προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος να ε, ε, ανέλθει και στην κοινότητα και στην κοινωνία ευνοεί πρώτα την εκμάθηση και στη συνέχεια τη χρήση γλωσσών που χαρακτηρίζονται σούπερ κεντρικές ή υπερκεντρικές. Και πέρα από την πολιτική ορθότητα και τα ωραία λόγια και τις ομιλίες για την πολυγλωσία και την προώθησή της και πέρα από την προώθηση της πολυγλωσίας γενικότερα υπάρχει αυτή η κατάσταση η οποία εξελίσσεται και εξελίσσεται διαβρώνοντας την γλωσσική ποικιλομορφία. Είτε χάνονται λοιπόν οι γλώσσες αυτές είτε περιορίζονται στην έκφρασή τους ή ακόμα και στο χώρο που ονομάζεται χώρος λειτουργικός μιας γλώσσας ε, και ε, χρησιμοποιούνται μόνο για ορισμένες δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής, ενώ από κάποιες άλλες αποκλείονται, διότι έχουν ε, αντικατασταθεί από υπερκεντρικές ή σούπερκεντρικές γλώσσες. Αυτή η δυναμική βεβαίως που οδηγεί οι ομιλούντες αυτές τις περιφερειακές γλώσσες τις μιλούν λιγότερο όταν βρίσκονται σε κάποιες δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής. Και μάλιστα πολλές φορές δεν τις μεταδίδουν τις γλώσσες αυτές στα παιδιά τους. Και ταυτόχρονα η ελίτ που ομιλούν αυτές τις γλώσσες, τις περιφερειακές και τις κεντρικές, συντονίζονται, συνεργάζονται ε, στις ε, σούπερ κεντρικές ή στην υπερκεντρική γλώσσα τα αγγλικά. Όπως είπε και ο κύριος Μαρτίνες προηγουμένως, ομιλούν έτσι μία γλώσσα που όχι μόνο δεν ομιλείται γενικότερα, αλλά δεν είναι κατανοητή από ε, ένα τμήμα ή ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ίδιου του του λαού ανεξάρτητα από τις όποιες προσπάθειες ε, εκμάθησης και ομιλώ με τα λόγου γνώσεως εδώ και ενώπιόν σας, ε, που ε, κάνουν οι κοινωνίες προσπάθειες για να διαδώσουν την πολυγνωσία και όχι μόνο οι κοινωνίες και οι μεγάλοι θεσμοί και μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε τις συστάσεις και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη για να διαδίδουν την πολυγνωσία. Ε, γνωρίζουμε όλα τα προγράμματα και όλες τις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένα εκεί. Και όλοι είμαστε διάπηροι υποστηρικτές ε, προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς ε, στη διακυβερνητική και ε, πολυμερή συνεργασία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι λιγότερο ευνοημένες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες αυτές η πολύγλωση εκπαίδευση είναι πολυτέλεια διότι αυτές οι χώρες έχουν την πρόκληση του να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό τους, όχι σε πολλές γλώσσες και έχουμε επαφές με προσώπους τέτοιων εκπαιδευτικών συστημάτων ε, χωρών, μας λέγουν ότι η πολυγλωσία στην εκπαίδευση είναι ωραία και ισχύει και εύκολη για τις χώρες του Βορρά, για κοινωνίες ε, προνομιούχες. Αλλά εμείς, αν, μπορούσαμε, ε, αν μπορούμε να πληρώνουμε τους δασκάλους μας, να μην έχουμε υπερβολικό αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη για να μπορούν να συγκεντρώνονται και να λειτουργούν σωστά, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Και πολύ συχνά εκπρόσωποι αυτών των κοινωνιών ανήκουν σε κοινότητε που είναι ήδη πολύγλωσσες. Από τη φύση τους, έτσι, την κοινωνική, όχι λόγω μόρφωσης. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτή η δυναμική οδηγεί σε μια χαλάρωση του γλωσσικού ιστού, σε μια απώλεια της λειτουργίας ορισμένων γλωσσών, κεντρικών αλλά και σούπερ κεντρικών και τελικά οδηγεί σε μια κοινωνιοπολιτική διάσταση, κοινωνικοπολιτική διάσταση. Υπάρχει ένα χάσμα δημοκρατικό ουσιαστικά. Ε, από τη μια έχουμε τις ελίτ που μιλούν αυτές τις γλώσσες, την υπερκεντρική και τις σούπερ γλώσσες και τις υπόλοιπες ή τους υπολείπους στη χώρα. Και όπως είπε ο κύριος Μαρτίνεθ εδώ όλοι μας και εσείς βεβαίως από τα εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά σας ε, καθήκοντα έχουμε μια βαριά ε, δημοκρατική ευθύνη και κατά κύριο λόγο και πρώτο το Κοινοβούλιο και αυτή η κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι μας όσοι εργάζονται στο θέμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσει κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους λαούς της Ευρώπης. Το είπε ο κ. Μαρτίνες, βρισκόμαστε σήμερα σε μια κρίση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και δύσκολο να ξεπεραστεί και ε, επιδεινώνεται η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλη την προστασία που προσπαθεί να οικοδομήσει. Φανταστείτε λοιπόν πώς φαντάζονται την Ευρώπη οι πολίτες μας όταν επιπλέον δεν κατανοούν τα όσα διαμείβονται, τα όσα λέγονται. Είναι ακόμα μεγαλύτερη η ματέωση εκείνων που δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να μιλήσουν. Και αναγκαστικά συνδέουν ε, αυτές τις καταστάσεις με αρνητικούς συνειρμούς στο μυαλό τους. Δεν μπορούν να έχουν θετική εικόνα από κάτι που δεν γνωρίζουν, που δεν κατανοούν και συχνά ε, όταν αγνοείς κάτι ή ε, δεν το γνωρίζεις αρκετά, δεν το εμπιστεύεσαι. Και έρχεται η καχυποψία. Αυτό ισχύει και για άλλους τομείς, ε, πέρα από την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, όπου οι λαοί απλούστατα είναι απόντες από τη δημόσια συζήτηση. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική συνέχεια, ένα σύνολο που έχουμε από τη μια της ελίτ, εδώ είμαστε μεταξύ πανεπιστημιακών και βουλευτών. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουμε μια ξύλινη γλώσσα διπλωματική ή γραφειοκρατική. Ε, οι ελίτ λοιπόν συνιστούν μια ουσιαστική ολιγαρχία. Και η συζήτηση γίνεται μεταξύ αυτών, σε μια γλώσσα που την κατέχουν εκείνοι, που μπορεί να είναι σούπερ κεντρική ή κεντρική, αλλά που ε, ζουν στον κόσμο τους ουσιαστικά. Και τους φαίνονται προφανή ε, κάποια πράγματα και κάποιες αποφάσεις και ε, δυσανασχετούν γιατί οι λαοί όχι μόνο δεν καταλαβαίνουν αλλά καμιά φορά απορρίπτουν στη δημοκρατική διαδικασία αυτές τις αποφάσεις. Και από την άλλη είναι αυτοί οι λαοί που ε, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, που έχουν την αίσθηση ότι είναι στο περιθώριο, παραγωνισμένοι και καμιά φορά όμως μπορεί να είναι και εκπρόσωποι και αιρετοί της κοινωνίας τους. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αλλού που σε διπλωματικά φόρα, σε κοινοτικά, όπως εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, μπορεί και πανεπιστήμια, επιχειρηματική κύκλοι, οποιοδήποτε σύνολο ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, όπου κυριαρχούν και χρησιμοποιούνται πάντα αυτές οι ίδιες γλώσσες. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πώς οδηγεί στις κοινωνίες, σε ένα δίλημα, μια πρόκληση και σε μια κατάσταση διπλής διαλεκτικής που είναι αρκετά περίεργη στο χειρισμό. Δηλαδή, είναι μια οργάνωση πολιτισμού που, ε, που εμπλουτίζει μάλλον την κοινωνία αφενός, αλλά από την άλλη ε, φτωχαίνει και από πλευράς πολυγλωσσίας και γλωσσικής και σε τελική ανάλυση δημοκρατίας. Ο εξορθολογισμός λοιπόν ορισμένων διαδικασιών, συστημάτων δημιουργεί φαινόμενα κυριαρχίας που αποκλείει τελικά ορισμένους. Ε, αυτή η δυναμική της παγκοσμιοποίησης ε, φέρνει τον κόσμο πιο κοντά, αλλά ταυτόχρονα ε, προκαλεί και αποκλεισμό, αλλά και κάποιες αγγυλώσεις ε, και περιχαράκωση ως προς την ταυτότητα. Και το βλέπουμε αυτό και στην κοινωνία μας. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα με αγωνίες, με φόβους, με ματέωση, με απογοήτευση απέναντι σε συζητήσεις που δεν κατανοεί ο κόσμος. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, οργανισμοί όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια κράτη ε, υιοθετούν γλωσσικές πολιτικές. Αυτές οι γλωσσικές πολιτικές αφορούν ε, κάποιες ρυθμίσεις για το καθεστώς των γλωσσών. Για, ε, αφορούν τις ίδιες τις γλώσσες, ας πούμε, μεταρρυθμίσεις γλωσσικές. Αφορούν επίσης καθεστώτα διερμηνίας, μετάφρασης. sur la transmission. Και για τη μετάδοση, πώς γίνεται αυτή με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση και βεβαίως και με το θέμα που μας ε, ενδιαφέρει σήμερα και με κάποια ε, χρήση των νέων τεχνολογιών να μπορεί κανείς να βοηθήσει και όχι να υποκαταστήσει τους διερμηνείς, τους μεταφραστές, είναι ένα υποβοηθητικό εργαλείο για το μέλλον. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει μια επιλογή. Και όπως είπε και ο κύριος Μαρτίνης, δεν είναι καθόλου αθώα αυτή η επιλογή, ούτε τυχαία. Είναι προϊόν πολιτικής βούλησης. Επελέγει λοιπόν το καθεστώς της πλήρους δερμηνίας. Ο καθένας ακούει τη γλώσσα του και έχει πρόσβαση μέσω της γλώσσας του στη διερμηνία και στη μετάφραση. Και ο καθένας μπορεί να επιλέξει να μιλήσει στη γλώσσα του, όπως έκανε ο κ. Μαρτίνες, και να τον, ερμηνεύουν, να τον διερμηνεύσουν επαγγελματίες που είναι και γλωσσομαθείς, αλλά πέρα ε, από τη γνώση αυτής καθ' του φορέα που είναι η γλώσσα, ε, είναι και άνθρωποι που περνάνε μηνύματα. Είναι πολιτιστικές γέφυρες Ακούσαμε για ενιδρίο εδώ. Αλλά μπορεί να είναι τελικά η σωστή μεταφορά, διότι σε αυτά τα ενιδρία έχουμε καταπληκτικά ψάρια που ελίσσονται ε, ε, πολύ άνετα ε, ανάμεσα στις, διάφορους πολιτισμούς. Εκεί που κάποιοι άλλοι είναι πιο άκαμπτοι και κανονικά θα έπρεπε να έχουν τη στοιχειώδη σύνεση, ε, να μην βουτήξουν στα βαθιά νερά. Αυτή λοιπόν η διαδικασία τελικά ενθάρρυνσης της πολυγνωσίας είναι ε, πολύ σημαντική. Δεν θα επιμείνω, είμαι στο συμπέρασμα, διότι δεν χρειάζεται να σας πείσω, το γνωρίζετε όλοι. Είναι σαφές ότι όσο περισσότερο αναπτύξουμε την πολυγνωσία και την εκπαίδευση και την κατάρτιση της γλώσσας αφές, τόσο περισσότερο θα δημιουργήσουμε ε, στην εκμάθηση της γλώσσας αυτή τη θαυμάσια ε, έννοια που είναι το να έρθει στη θέση του άλλου ή το να της μεταβολής. Δηλαδή, άλλο είναι η ετερότητα και άλλο είναι το να μπει ε, στη θέση του άλλου. Και έχουμε ανάγκη την ανεκτικότητα και την ανοχή και όχι να δυσπιστούμε και να είμαστε καχύποπτοι απέναντι στον άλλο, απέναντι στον έτερο, αλλά να έχουμε περιέργεια. Και εκείνοι που έχουν ε, την ε, ε τύχη, τη χάρη να είναι πολύγλωσσοι, γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θαυμάσιο χαρακτηριστικό, δείχνει ανοιχτό πνεύμα και δυνατότητα να μπορεί κανείς να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του άλλου. Και ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ περίπλοκο, όπου όταν βλέπεις τον κόσμο μέσα από ένα και μοναδικό φίλτρο είναι πολύ μεγάλη φτώχεια. Ο πλούτος του κόσμου είναι τέτοιος που χρειαζόμαστε όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες να δούμε τον κόσμο από διαφορετική σκοπιά. Και κάθε γλώσσα είναι ένα μετερίζει από όπου βλέπεις τον κόσμο και την οργάνωσή του με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό είναι σαφές ότι έτσι μπορούμε να αλλάξουμε κιόλα. Γιατί όταν ανταλλάσσουμε σημαίνει ότι αλλάζουμε και οι ίδιοι. Και η βάση αυτών είναι η γλώσσα. Όσο περισσότερες γλώσσες μαθαίνουμε, όσο περισσότερες γλώσσες μιλάμε, τόσο πιο ανοιχτοί είμαστε απέναντι στους άλλους. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας, γιατί πρέπει να το πω αυτό, με κάτι ρεαλιστικό. Σας μίλησα για τη διάβρωση ε, της ε, γλωσσικής ποικιλομορφίας. Αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα και πρόσφατες μελέτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωβαρόμετρο Φερρυπίν του 2012, δείχνουν ότι όλοι είναι πεπισμένοι για την ευεργετική επίδραση της πολυγλωσσίας και οι ίδιοι λαοί, αλλά παρόλα αυτά τι διαπιστώνουμε μειώνεται η γλωσσομάθεια και υπάρχει και ανασφάλεια γλωσσικών, ε, γλωσσο, ε, εκείνων που μιλούν μια γλώσσα. Δηλαδή όχι μόνο ο κόσμος μιλάει λιγότερες γλώσσες, αλλά και όταν τις μιλάει θεωρεί ότι δεν τις μιλάει αρκετά καλά. Και τη μόνη γλώσσα που θεωρεί ο καθένας ότι τη μιλάει πάνω κάτω καλά είναι αυτή η υπερκεντρική όπως είπαμε. Επειδή έχω πολύ ταξιδέψει ε, και ακούσει πολλά και ζήσει, επιτρέψτε μου λίγο να αμφιβάλλω. Απομένουν βεβαίως να γίνουν πολλά ε, για να πιστούν οι λαοί και οι φοιτητές, προκειμένου που είναι το μέλλον των λαών, για την ανάγκη να μαθαίνουν νέες γλώσσες, να εκπαιδεύονται. Επίσης πολλά απομένουν για να πιστούν όλοι, συμπεριλαμβανομένων δε και των ε, μελών αυτών των ελίτ, ότι θα πρέπει να εμπιστεύονται τους διερμηνείς περισσότερο από τον εαυτό τους. Ότι θα πρέπει να σέβονται τους λαούς από τους οποίους προέρχονται και στους οποίους ανήκουν, μιλώντας τη γλώσσα της δικής τους ταυτότητας, την οποία είναι βέβαιη ότι θα εκφραστούν καλύτερα από ό,τι όταν μιλούν άλλες γλώσσες. Και να αφήσουν στους επαγγελματίες διερμηνείς να κάνουν τη δουλειά αυτή να δημιουργήσουν τη γέφυρα και το σύνδεσμο με τις άλλες κουλτούρες και τους άλλους πολιτισμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μεταφράζει κανείς, δεν ε, διερμηνεύει μόνο. Είναι πολύ περισσότερο. Είναι ένα σύνδεσμος μεταξύ των πολιτισμών και αυτός είναι ο ρόλος και το επάγγελμα των διερμηνέων. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η εκπαίδευση, κατάρτιση και ίσως οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν και μπορούν να συνεισφέρουν ε, ουσιαστικά Ήθε οι εργασίες μας να ακολουθήσουν αυτή την ατραπό στη μεγάλη παράδοση που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε κύριε Λοπέζ. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ε, θα σας δώσω το λόγο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Λοπέζ ε, σε σχέση με την στάση των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε σχέση με την πολυγλωσία. Διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέβεται απόλυτα την πολυγλωσία με τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ βλέπω πως υπάρχουν μόνο 9 ε, γλώσσες μετάφρασης, συνήθως υπάρχουν 23. Α, όχι, είναι πάνω, δεν τις έχει δύο μιλητές στις υπόλοιπες γλώσσες. Καλά να πάθω, είναι διόροφες οι καμπίνες. ναι, διόροφο το ενιδρίο. Δεν το είχα αντιληφθεί. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γλώσσες εργασίας. Και ήθελα να επιμείνω για το γεγονός ότι η έλλειψη πολυγλωσσίας δημιουργεί μια ε, δυσπιστία και καχυποψία, αυτή εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο απέναντι στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο ή μήπω θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι το Κοινοβούλιο βγαίνει σχετικά ανέπαφο από αυτή τη διαδικασία, στη σχέση δηλαδή με του Ευρωπαίου πολίτε, γιατί το Κοινοβούλιο σέβεται απόλυτα την πολυγλωσία. Φυσικά αυτό το πρόβλημα καχυποψίας αφορά περισσότερο, στρέφεται μάλλον περισσότερο κατά τη Κομισιόν. Δεν θέλω να είμαι πολιτικό ε, λάθος, αλλά υπάρχουν αποχρώσει σε αυτή την αντίληψη. Να απαντήσω ότι είναι ε, η ίδια η φύση του Κοινοβουλίου σχέση του με τους λαούς να επαγρυπνεί ε, όσον αφορά το θέμα της πολυγλωσσίας, διότι ένας βουλευτής που εκλέγεται δεν μπορεί εύκολα να καταργήσει τη γλώσσα του λαού του. Θα του κοστίσει πολύ ακριβά κάτι τέτοιο. Ούτε η δουλειά του βουλευτή δεν είναι εύκολη, αλλά αν ξεχνάγε και τη γλώσσα του λαού που τον εκλέγει, θα είχε σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό και το Κοινοβούλιο επαγρυπνή δεν είναι μόνο η πρωτοβουλία των βουλευτών, Υπάρχει η βούληση του Κοινοβουλίου να φροντίζει ιδιαίτερα το θέμα της πολυγλωσσίας είναι ένα θεσμικό όργανο υποδειγματικό από αυτή την άποψη. Η Κομισιόν βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Από τη φύση της δεν είναι μέσα στον δημοκρατικό λόγο και συζήτηση έχει πολύ τεχνικές και πρακτικές αρμοδιότητες. Ε, ε, εκείνη αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες για τα διάφορα θέματα για να προχωρήσει η Ένωση και στην ουσία αυτό που με εντυπωσιάζει όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, εμένα με εντυπωσιάζει αυτή η ταχύτητα. Μα πολλοί λένε ότι προχωράει πολύ αργά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εγώ πιστεύω πως αντίθετα είναι μια, ένας αγώνας δρόμου και η δυσκολία της Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο βέβαια έχει να κάνει πολλά ταυτόχρονα, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει κανείς να είναι γρήγορος, αποτελεσματικός και να αντιδρά γρήγορα στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά πρέπει απόλυτα να γίνεται σεβαστή η ακρίβεια καταρχήν, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι εξαιρετικά περίπλοκες συζητήσεις όπως αυτές που γίνονται στην Κομισιόν μπορούν πάντοτε να γίνονται σε γλώσσες που δεν ε, τις ε, κατέχει απόλυτα καλά ο κάθε ομιλητής. Και εγώ ε, θα μπορούσα να σας μιλήσω στα γερμανικά, για παράδειγμα, ή στα αγγλικά, αλλά δεν το έκανα. Διάλεξα τη γλώσσα μου, τη μητρική μου γλώσσα και το έκανα επίτηδες. Ε, νομίζω λοιπόν πως και η Κομισιόν έχει να αντιμετωπίσει μια πρόκληση, γιατί είναι γεγονός ότι η πολυγλωσία μειώνεται. Ωστόσο, θα ήθελα να κλείσω λέγοντα το εξή. Και εγώ πιστεύω στην ατομική ευθύνη. Και εγώ ανήκω σε έναν πολυμερή οργανισμό που είναι η Διεθνή Οργάνωση τη ε, ε, Γαλλομάθειας. Ε, έχουμε 27 χώρε. Δεν μπορούμε διαρκώ να κατηγορούμε του θεσμού ότι αυτέ φταίνε. Αυτή, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη, είναι 27 κράτη. Βούληση σε αυτά εναπόκειται. Οι θεσμοί αποτελούνται από τα κράτη. Και άρα λοιπόν αυτά τα κράτη έχουν εκπροσώπους που δεν πάβουν να φέρουν την ταυτότητά τους από τη στιγμή που μπαίνουν σε ένα διεθνές όργανο. Δεν αφήνουν πίσω τους την ταυτότητά τους στη, στην, στους αλάμους ασφάλειας έχουν, φέρουν την ευθύνη και τη γλωσσική τους ταυτότητα να την έχουν μαζί τους. Γιατί αυτή είναι η φορή αυτής της διαφορετικότητας, της πολυμορφίας, της πολιτιστικής. Είναι ευθύνη του καθενός. Και εδώ πιστεύω πως μπορεί εσείς όντως να έχετε την ευθύνη ως ε, μεταβιβαστές γνώσης και εμπειρίες να ευαισθητοποιήσετε τους φοιτητές δεν είναι δυνατόν η γλωσσική συνείδηση να είναι μόνο προτεραιότητα εν μειονών κάποιων κοινωνιών που είναι σε μειονότητα στην ουσία γλωσσικά. Θα έπρεπε ο καθένας να έχει τη συνείδηση ότι φέρει, ε, ο ίδιος είναι φορέας ενός πολιτιστικού και γλωσσικού κληροδοτήματος και δεν πρέπει να το εγκαταλείπει τυχοδιοκτικά ε, ελαφριά την καρδιά. Η Κομισιόν δεν μπορεί βέβαια να, με το βούρδουλα πίσω από κάθε, πάνω από το κεφάλι κάθε υπαλλήλου να τον υποχρεώνει να μιλά τη τάδε δίνα γλώσσα. Όχι, είναι και ατομική ευθύνη του καθενός. Αυτά, ευχαριστώ. Μάλιστα, θέλει κανείς να θέσει μια ερώτηση. Μάλιστα, κύριε Μπενεντέτη. Ονομάζομαι Μάρκο Μπενετέτη και είμαι Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Διερμηνίας της Κομισιόν, εφόσον γίνεται λόγος για αυτήν. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να παρέμβω για αυτό το σημείο. Εγώ ε, συμφωνώ με το όσο είπε ο κύριος Λοπές, εκτός από το εξή ότι η δυσκολία των συζητήσεων είναι εμπόδιο στην πολυγλωσία. Δεν πιστεύω πως οι διερμηνείς μας δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε δυσκολία. Το πράττουν αυτό καθημερινά. Αντίθετα, είναι αλήθεια ότι η φύση, η ταχύτητα, η ένταση και ο αριθμός των συνεδριάσεων της Κομισιόν και ε, στην ουσία η έλλειψη διερμηνέων σε ολόκληρο τον κόσμο να μην επιτρέπει να καλύπτονται από πλήρη γλωσσικά καθεστώτα όλες τις συνεδριάσεις της ε, Κομισιόν. Ωστόσο, η υπηρεσία την οποία εγώ διευθύνω εξασφαλίζει τη διερμηνία και στις, ε, για τις συνεδριάσεις των Υπουργών, του Συμβουλίου των Υπουργών. Και εκεί γίνονται σε όλες τις γλώσσες, διότι πρόκειται για την ίδια δημοκρατική συζήτηση που γίνεται εκεί για το ίδιο επίπεδο εκπροσώπησης. Άρα λοιπόν, ίσω στην Κομισιόν να μην είμαστε τόσο γλωσσοί όσο στο Κοινοβούλιο, αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίε διερμηνία τη Κομισιόν έχουν, και εγώ πρώτο και καλύτερο, φροντίζουν την ποιότητα της πολυγλωσσίας και τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Και για μας λοιπόν η πολυγλωσία είναι προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση κύριε Γενική Διευθύντα. Υπάρχει κάποιος άλλος να θέλει να πάρει το λόγο. Εφόσον όχι, Ίσως μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι. Πιστεύω πως είμαστε μέσα στα χρονικά όρια που από την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καϊλά και κύριε Λόπες. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τώρα πριν βγείτε όλοι έξω γιατί έχουμε διάλειμμα για καφέ όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Αλλά παρακαλώ να ξαναγυρίσετε. Αξίζει τον κόπο στις 4.30 γιατί θα ε, μπούμε σε μια σημαντική ενότητα για τα πανεπιστήμια, δυνατότητες χρηματοδότησης για προγράμματα κινητικότητας και άλλα πράγματα. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να ξαναγυρίσετε στην ώρα σας. Θα κάνουμε και μια μικρή οικογενειακή φωτογραφία τώρα στο διάλειμμα, γιατί δεν τα κάνει μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτά και εμείς. Και αν θέλετε ένα password για το ασύρματο διαδίκτυο, ε, ρωτήστε έξω στη γραμματεία και για τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα το διαθεσμικό ε, για επιδοτήσεις πανεπιστημίων απευθυνθείτε στο συνεργάτη μου, τον κύριο Εμίλιο Ορλάντο και μπορείτε να του κάνετε και τις πρακτικές σας ερωτήσεις και με χαρά ε, θα σας απαντήσει. Λοιπόν, καλό σας διάλειμμα και ευχαριστώ και πάλι. I would like to welcome you back to this session uh, Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δεύτερο πάνελ που αφορά το αέρασμα στην κινητικότητα και τα κοινά προγράμματα σπουδών Αν Άμα επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα τουρκικά, και να αφήσω τους συναδέλφους ε, να με μεταφράσουν ε, με την επιδειξιότητα που του χαρακτηρίζει στις δικές τους μητρικές γλώσσες. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο πάνελ. Θα πρέπει τώρα, όπως προβλέπει και ο τίτλος, να συζητήσουμε για το Erasmus Mundus, το πρόγραμμα ανταλλαγών με τα πανεπιστήμια, που είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα αυτά τα κοινά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για τα πανεπιστήμια και φυσικά και το χρηματοοικονομικό του σκέλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια τα οικονομικά ζητήματα σε όλους τους τομείς είναι ενδιαφέροντα, είτε αφορούν το Εράσμος, είτε αφορούν άλλα προγράμματα. Σίγουρα η χρηματοοικονομική πτυχή αποτελεί σημαντικό σκέλος των προγραμμάτων. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αφιερώσει ένα τμήμα του σεμιναρίου στο πρόγραμμα αυτό. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα μέλη του πάνελ. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι πολύ σημαντικό για μα. Είναι ο κύριο Βίτο Μπορέλη, ο αρμόδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Ο κύριο Μπορέλη είναι επιφορτισμένος με την επίλυση των προβλημάτων του Erasmus Mundus και με ιδιαίτερη χαρά του δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ και του συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με προσκάλεσαν για να σας παρουσιάσω σήμερα το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Ε, αισθάνομαι κάποια μηχανία και τρακ ε, που λαμβάνω το λόγο μετά τους ε, πολύ τους, τις ομιλίες που χαρακτηρίζονται από μεγάλο ίστρο αλλά και πολιτική αυθεντία και κύρος και επίση αισθάνομαι και μηχανία γιατί είμαι Ιταλός και σήμερα θα σας μιλήσω αγγλικά αλλά εκπροσωπώ εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρθηκε πολλές φορές ως θεσμικό όργανο που δεν είναι και πολύ φιλικό προς την πολυγλωσία. Και ε, οφείλω να ομολογήσω ότι στις περισσότερες μας συνεδριάσεις χρησιμοποιούμε λίγες γλώσσες εργασίας για να μην πω μία και μόνο γλώσσα εργασίας. Και δεν χρειάζεται να σας διευκρινίσω ποια. Σα ζητώ συγγνώμη λοιπόν που μιλώ αγγλικά, αλλά αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιούμε καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πραγματευόμαστε τέτοια θέματα, δηλαδή πανεπιστημιακή συνεργασία ε, και κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών. Το θέμα της σημερινής ε, διάσκεψης είναι οι νέες τεχνολογίες ε, και η παιδεία για την πολυγλωσία. Και σίγουρα το πρόγραμμα Erasmus Mundus ε, έχει πολύ στενούς και ισχυρούς δεσμούς με αυτό το θέμα. Γιατί παρά τις γνωστές και ευρύτερες επικρίσεις που ακούγονται πολλές φορές για την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση εξαιτία της ε, ομοιογενοποίησης που τη χαρακτηρίζει ως προς την γλώσσα διδασκαλία που είναι τα αγγλικά. Με ιδιαίτερη χαρά οφείλω να πω ότι το πρόγραμμα Erasmus Mundus από την αρχή του προώθησε την ε, πολυγλωσία και τη χρήση των εθνικών γλωσσών, αν όχι για λόγους διδασκαλίας, τουλάχιστον ως υποχρεωτικό θέμα του προγράμματος σπουδών που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών, ιδιαίτερα ε, των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ε, μεταπτυχιακών και διδακτορικών του Erasmus Mundus, ομολογώ ότι δεν είναι και πολλά αυτά τα προγράμματα σε θέματα γλωσσών. Και από ό,τι θα γνωρίζετε και οι περισσότεροι από εσά, αυτό οφείλεται στο ότι κατά παράδοση η πανεπιστημιακή συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο ήταν πιο α, συχνή σε θέματα κοινωνικών επιστημών, φυσικών επιστημών και ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των μαθημάτων μας αφορούν ανθρωπιστικές σπουδές. Και σε αυτό το μικρό ποσοστό, ένα ακόμη πιο μικρό ποσοστό, αφορούν τις γλώσσες. Βέβαια, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, η εκμάθηση γλωσσών, η μελέτη γλωσσών δεν είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό ε, των πανεπιστημίων για συνεργασία. Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα κοινή ε, ανάπτυξη με πολλέ χώρε ε, προγραμμάτων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών στο τομέα της πολυγλωσία, ε, που είναι μέσο για κοινωνική ανάπτυξη ή για την ανάδειξη τη σημασία κάποιων περιφερειακών γλωσσών, γλώσσων μειονοτήτων ή τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών και τη χρήση τους στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στη διερμηνία. Όφελα να κάνω αυτή την εισαγωγή για να δώσω και το πλαίσιο της ε, σημερινής μου παρουσίασης που θα εστιαστεί κυρίως στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Πριν όμως σας ε, εξηγήσω τις διάφορες δράσεις του προγράμματος αυτού, θα ήθελα εν συντομία να σας υπενθυμίσω τους πολιτικούς στόχους του προγράμματος Erasmus Mundus, που είναι πάνω κάτω οι ίδιοι από την ε, έναρξη του προγράμματος το 2004. Το πρόγραμμα λειτουργεί πια εδώ και 8 χρόνια και η στόχη του είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτερης Εκπαίδευσης μέσω της διεθνούς συνεργασίας και αυτό γίνεται με την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών προγραμμάτων που εκπονούνται από ομάδες ε, Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την πιθανότητα να, να συμπεριληφθούν στα προγράμματα αυτά και εξοκοινοτικοί εταίροι. Δεύτερος στόχος του Ερασμούς Μούντους είναι η βελτίωση της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων. Πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα μέσω της ε, μεγάλης κρίσης και της ανεργίας. Είναι σημαντική ανώτερη εκπαίδευση γιατί δίνει περισσότερα εφόδια και επαγγελματικές ευκαιρίες στους φοιτητές. Και περνάμε τώρα σε ένα πιο πολιτικό στόχο του Erasmus Mundus που είναι η πρόθεση του διαλόγου και της κατανόησης ε, και συνεννόησης μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και να διδάσκουμε γλώσσες ε, και τον πολιτισμό. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορούν να προσφέρουν τα πανεπιστήμια στους φοιτητές τους. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα Erasmus Mundus απευθύνεται κυρίως σε εξοκοινοτικούς φοιτητές που έρχονται να σπουδάσουν στην Ευρώπη, τουλάχιστον ε, ένα τμήμα των σπουδών τους, να το παρακολουθήσουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Οπότε τέταρτος στόχος του Erasmus Mundus είναι η πρόθεση της Ευρώπης ως κέντρο αριστείας ε, της γνώσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή θέλουμε να καταστήσουμε τη δική μας ανώτερη εκπαίδευση πιο ελκυστική, πιο διαφανή, αλλά και πιο ανταγωνιστική απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να σας παρουσιάσω την δομή του προγράμματος Erasmus Mundus. Η δομή αυτή πέρασε από διάφορες φάσεις. Η πρώτη ήταν το 2004-2008 και η δεύτερη φάση είναι αυτή που διανύουμε σήμερα, 2009-2013. Περιμένουμε να συνεχιστεί το πρόγραμμα και μετά το 2014. Η πρόταση όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα που θα το διαδεχτεί λέγεται Erasmus for All, Erasmus για όλους και θα είναι ένα πρόγραμμα πλαίσιο στο οποίο θα συμμετέχουν όχι μόνο το Erasmus Mundus αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus, Leonardo da Vinci, το πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Θα πρόκειται για ένα πρόγραμμα γενικό που θα καλύπτει πολλά επιμέρους προγράμματα και θα περιλαμβάνει και τις δραστηριότητε που σήμερα εντάσσονται στο Erasmus Mundus. Η πρώτη δράση είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματος, γιατί προωθεί την συνεργασία πανεπιστημίων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών και το συνδυάζει με ε, υποτροφίες που όπως είπα δίνονται κυρίως σε εξοκοινοτικούς φοιτητές για να σπουδάσουν στην Ευρώπη και σε εξοκοινωτικούς ε, καθηγητές που συνεχίζουν τη διδασκαλία και τις ερευνητικές του δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από το 2009 χρηματοδοτεί υποτροφίες και για Ευρωπαίους φοιτητές. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι το βασικό στοιχείο του προγράμματος. Γιατί οι υποτροφίες για Ευρωπαίους είναι λιγότερες από τις υποτροφίες που δίνουμε σε έξω φοιτητέ. φοιτητές. Η δεύτερη δράση του προγράμματος στηρίζεται σε συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, αλλά στόχος δεν είναι η ανάπτυξη κοινών ε, προγραμμάτων σπουδών και πτυχίων, αλλά ε, δημιουργία μιας, πλατφόρμα πλατφόρμας φοιτητών. Επικεντρώνεται δηλαδή σε βραχυπρόθεσμη κινητικότητα, και όχι κινητικότητα σε προπτυχιακό επίπεδο που εμπίπτει περισσότερο στην πρώτη δράση ή σε μεταπτυχιακό. Και η τρίτη δράση είναι κάποια προγράμματα προώθησης, σχέδια προώθησης, που δεν εφαρμόζονται κατά ανάγκη από πανεπιστήμια μόνο, αλλά και από διάφορους φορείς προώθησης ε, της εκπαίδευσης ή από άλλους διεθνείς φορείς ε, που ε, ενισχύουν την συνεργασία στην ανώτερη εκπαίδευση. Μπορεί να πρόκειται για σχέδια, ε, προγράμματα, μελέτες, ε, έρευνες, φεστιβάλ, εκθέσεις και ε, στόχο τους έχουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανώτερη εκπαίδευσης εν ώψη τη Και κάποια στοιχεία για να δείτε την ευέλεια του προγράμματος. Μέσα στην οκταετή εφαρμογή του, το πρόγραμμα Erasmus Mundus έχει υποστηρίξει περίπου 150 κοινά μαθήματα μεταπτυχιακών 50 κοινά προγράμματα διδακτορικών σπουδών, 50 εταιρικέ σχέσει ε, τύπου δράση 2 για ανταλλαγή φοιτητών και 60 σχέδια προώθηση ε, τη της, ε, δράσης 3. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι υποτροφίες και την κινητικότητα του προγράμματος. Στα κοινά προγράμματα που έχουμε στα πλαίσια της πρώτης δράσης, μέσα στην οκταετία δώσαμε υποτροφή σε πάνω από 15.000 φοιτητέ και μεταπτυχιακούς ε, και σε πάνω από 2.000 καθηγητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού. Επίσης, ε, στη δεύτερη δράση, σε πάνω από 25.000 φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού και μάλιστα ε, το, το, το αριθμός είναι υψηλότερος γιατί είναι πιο βραχυπρόθεσμες η δράση και η παραμονή. Και μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2013 αναμένεται ότι θα φτάσουμε στους 50.000 συνολικά φοιτητέ και καθηγητές που θα υποφελούνται από το πρόγραμμα. Τώρα, για να σας δώσω μια ιδέα για τις πιο δραστήριες χώρες του προγράμματος, η πρώτη χώρα είναι η Ινδία για υποτροφίες σε φοιτητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες για την πανεπιστημιακή συνεργασία η Κίνα είναι δεύτερη και για τις δύο κατηγορίες, ιδιαίτερα δραστήρια λοιπόν. Η Κίνα και μερικές άλλες χώρες που παίζουν επίσης ρόλο, οι χώρες BRICS, αλλά και κάποιες αφρικανικές χώρες όπως η Αιθιοπία, που είναι πόρο η χώρα που στέλνει το μεγαλύτερο βαθμό υποψηφιωτήτων και αιτήσεων. Δεν είναι βέβαια η χώρα από τι οποίε επιλέγονται οι περισσότεροι φοιτητέ, αλλά σίγουρα είναι η χώρα την οποία υποβάλλονται οι περισσότερε αιτήσει υποτροφιών. Ίσως ε, επειδή τα πανεπιστήμια, η, Αιθιοπική, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Αιθιοπία είναι ιδιαίτερη, ιδιαίτερα δημοφιλής και αποτελεσματική στο έργο τους. Πάντως λαμβάνουμε πολλές αιτήσει από την Αιθιοπία. Και θα ολοκληρώσω με μερικές διαφάνειες που δείχνουν κάποιες ε, συμπληρωματικές δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus Mundus. Και επίσης να σας δείξω πόσο μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του προγράμματος. Οι διάφοροι αυτοί τομεί, τα κλάστερ του Erasmus Mundus, είναι μια πρωτοβουλία για να αξιοποιηθούν συνέργειε και να εντοπιστούν οι καλύτερε πρακτικέ στα διάφορα προγράμματα του Erasmus Mundus. Εντοπίσαμε πέντε τομεί για του οποίου θέλουμε ε, αξιοποίηση και ανταλλαγή των καλύτερων αποτελεσμάτων. Είναι η βιωσιμότητα, η απασχολησιμότητα, η αναγνώριση, ένα τομέα αφορούσε τα προγράμματα της Περιφερειακής Ασίας, δηλαδή συνεργασία ιδιαίτερα με πανεπιστήμια της Ασίας και ε, ένα θεματολογικό τομέα που ήταν οι κλιματικές αλλαγές. Βλέπετε και το link μας στην ιστοσελίδα. Η ΕΜΚΟΑ, η διασφάλιση ποιότητας των μαθημάτων, είναι κάτι που επίση εφαρμόζουμε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Γίνεται μια ανάλυση της ποιότητα των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μάστερ και δοκτορά, διδακτορικών. Επίσης έχουμε ένα εγχειρίδιο ποιότητας που δίνουμε οδηγίες σε τωρινούς και μελλοντικού ε, μετέχοντες του προγράμματος και ένα online εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση. Εκεί μπορούν να συγκρίνουν οι διάφοροι φοιτητέ ε, τις επιδόσεις τους με κάποια προκαθορισμένα κριτήρια αριστείας που έχουμε εκπονήσει στο Erasmus Mundus. Έχουμε και μία άλλη πρωτοβουλία για τους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Τους δίνουμε πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στα εθνικά, στις εθνικές ιστοσελίδες ε, και να βρουν πληροφορίες όχι μόνο για κοινοτικά προγράμματα όπως το Erasmus αλλά και για προγράμματα εθνικών υποτροφιών στις διάφορες χώρες μέλη. Και ένα από πιο επιτυχημένα σημεία και τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες του Erasmus Mundus είναι η δημιουργία ε, των ε, συλλόγων φοιτητών και αποφύτων του Erasmus Mundus με την πρόθεση δικτύωση και επαφών ε, και με άλλους εταίρους του δικτύου και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις πρωτοβουλίες της διεθνώς. Έχουμε μάλιστα σήμερα γύρω στους 7.000 φοιτητές και αποφύτους που συμμετέχουν σε, αυτή την, σε αυτό το σύλλογο και μάλιστα ε, είναι η πιο πιστική και σημαντική μας πρέσβησα ανά τον κόσμο. Γιατί αυτοί προβάλλουν το πρόγραμμα στον κόσμο και ελπίζουμε ότι οι φοιτητέ, αφού ολοκληρώσουν τι σπουδέ του στην Ευρώπη, θα επιστρέψουν στου πατρίδε και θα προωθήσουν, θα συνεχίσουν την πρόθεση και την προβολή τη Ευρώπη και στι δικέ του χώρε και θα δημιουργήσουν πολιτιστικού και άλλου οικονομικού δεσμού. Έχετε στι ιστοσελίδε αυτέ και πολύ πιο λεπτομεριακές πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσοχή και είμαι στη διάθεσή σας για να επιλύσω τις, απο... λύσω τις απορίες σας και να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλη. Εάν έχετε ερωτήσεις, κρατήστε τις για το τέλος ε, του πάνελ. Θα ακούσουμε πρώτα όλους τους ομιλητές και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στην κυρία Μπελέν Μπερνάντο Ντεκεϊρός. Είναι κάποια που γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια ήδη, διότι τη γνωρίζω από τα μαθήματα του Ζαν Μονέ και είχα διαρκώ επαφέ μαζί τη, στο και αν ήταν ανταλλαγέ ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αντιπροσωπεύει εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τη δώσω αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Εμπρού και εγώ χαίρομαι πολύ που σε βλέπω σήμερα και αν και έχω προετοιμάσει την ε, παρουσίασή μου στα αγγλικά και στα γαλλικά, γιατί εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν για την ε, Παιδεία και τον Πολιτισμό και είμαι και τμήματάρχης της ε, Μονάδας για την Πολυγλωσία. Θα μιλήσω στα Ισπανικά. Γιατί? Ε, γιατί αφού άκουσα την ομιλία του κυρίου Μαρτίνε, δεν μπορώ παρά να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα ως ένα φόρο τιμής προς τον ίδιο και τα λόγια του και το μήνυμά του που ήταν τόσο εμπνευσμένο και μας εμπνέει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς τους καιρούς που είναι τόσο χαλεποί της ιστορίας μας. Θα σας μιλήσω κυρίως για τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Πώς χρηματοδοτούμε εμείς λοιπόν τις γλώσσες στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Αυτό το καιρό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολυετές, από το 2007 μέχρι το 2013 είναι η προγραμματική περίοδος και είναι η διαβίου μάθηση. Ε, βλέπετε εδώ πόσο διαρκεί το πρόγραμμα, ποιες είναι οι βασικές ε, πληροφορίες για να μπείτε στην ιστοσελίδα και τη δομή του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαιρείται σε τέσσερα μεγάλα χρονολογικά προγράμματα. Κομένιους για το σχολείο, Εράσμος για το Πανεπιστήμιο, Λεωνάρδο για την κατάρτιση και ο Κρούντβικ για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Και έχουμε και δύο εγκάρσια προγράμματα που είναι το Ζωμονέ, όπως είπε η Εμπρού στην αρχή, που ε, αφορά τις σπουδέ για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένα άλλο εγκάρσιο πρόγραμμα που έχει διάφορες δράσεις τις οποίες επικεντρώνεται. Νέε τεχνολογίες είναι μία από αυτές. Άλλοι είναι οι γλώσσες. Και εδώ ε, βλέπουμε τη χρηματοδότηση στην οποία θα αναφερθώ. Το πρώτο που θέλω να σας αναφέρω είναι ποιες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Γιατί, διότι Πολλές από τις χώρες που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν παρευρίσκονται σήμερα με πριτάνεις και εξέχονται στις εκπροσώπους. Εκτός λοιπόν από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα φυσιολογικό, ε, μπορούν να συμμετέχουν, είναι επιλέξιμες δηλαδή, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που είναι Ισλανδία, Λίχτενστάιν και Νορβηγία, οι σκανδιναβικές χώρες και η Κροατία, η Τουρκία, η Ελβετία πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία. Γιατί γνωρίζω ότι παρευρίσκονται και εκπρόσωποι τους. Και τελευταίο, σύνολο είναι η Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Μαυροβούνιο. Μια μικρή διευκρίνηση. Η Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Μαυροβούνιο πρέπει ακόμα να ε, ε, πληρώσουν μια μικρή διατύπωση να υπογράψουν μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ολοκληρωθεί αυτή την πρώτη του μηνός ε, επιλογής ε, το επόμενο έτος, τότε όλα θα πάνε καλά. Αλλιώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι μείζον δυσκολία κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν στις γλώσσες και τα χρήματα που έχουμε και τι χρηματοδοτούμε. Στη δράση παριθμών 2 του προγράμματος του εγκαρσίου για τις γλώσσες έχουμε ένα προϋπολογισμό περιορισμένο, 10 εκατομμύρια μόνο για τις γλώσσες και πρέπει να σας πω ότι ο προϋπολογισμός που αφιερώνεται στις γλώσσες σε όλο το πρόγραμμα της διαβίου ε, μάθησης είναι πάνω από 50 εκατομμύρια συνολικά, γιατί κάθε ένα από τα τομεακά προγράμματα χρηματοδοτεί και γλώσσες. Αυτό όμως που μπορεί να σας ενδιαφέρει εσά για την πανεπιστημιακή συνεργασία είναι τα 10 εκατομμύρια λίγο περισσότερο από 7 πηγαίνει σε ε, πολυμερή προγράμματα που θα σας εξηγήσω ε, στη συνέχεια. Πάνω από 2 εκατομμύρια είναι τα δίκτυα και πάρα πολύ συμβολική ε, είναι η χρηματοδότηση των συνοδευτικών μέτρων. Θα σας παρακαλούσα να συγκρατήσετε το εξής από τη συγκεκριμένη διαφάνεια. Στα πολυμερή έργα που μπορεί να συμμετέχετε πολλοί από εσά, χρηματοδοτούμε μέχρι 200.000 το χρόνο. Αλλά επειδή τα προγράμματα μπορούν να είναι τριετή, ε, κατανοείτε ότι το, το μέγιστο, ε, η οροφή είναι 400.000, που 400.000 επιτρέπουν πολλά να γίνουν. Στα δίκτυα λοιπόν και τα συνοδευτικά μέσα, το μέγιστο κατέτος είναι 150.000. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στα πολυμερή ε, έργα και προγράμματα. Ε, μπορεί να τρέχει το πρόγραμμα τρία χρόνια, όπως και το δίκτυο, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί όλη η προσπάθεια. Ε, τα συνοδευτικά μέτρα είναι αιτήσια, η ενιάψια και το πιο σημαντικό είναι ο αριθμός των χωρών που θα πρέπει να συμμετέχουν για να είναι επιλέξιμο το πρόγραμμα. Στα ε, πολυμερή προγράμματα είναι τρεις χώρες, η μία θα πρέπει να είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ανοιχτή αυτή η δράση στον υπόλοιπο κόσμο. Το ίδιο ισχύει για τα δίκτυα και για τα ε, συνοδευτικά μέτρα είναι επιλέξιμη μόνο μία χώρα κάθε φορά. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι έχει ε, προκηρυχθεί, προσπαθευτεί και η επιλογή θα γίνει μετά το τέλος Φεβρουάριου λέγει η προθεσμία και τον Ιούλιο θα υπάρχουν τα αποτελέσματα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα έργα, τα πολυμερή. Δεν θέλω να σας διαβάσω τη διαφάνεια που βλέπετε. Δεν έχει νόημα άλλωστε. Είναι μια σύμπραξη ε, ε, φορεών που μπορεί να είναι πολιτιστικά Ινστιτούτα, πανεπιστήμια ή άλλοι φορείς που είτε ευαισθητοποιούν ε, για το θέμα των γλωσσών είτε ε, διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Μία από τις ε, πρωτοβουλίες που είναι πιο ισχυρές, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι τα περίφημα μαθήματα online, επιγραμμικά εκμάθησης γλωσσών. Νέες τεχνολογίες είναι και το θέμα που σας απασχολεί. Είναι πεποίθησή μας ότι βεβαίως τα μηχανήματα δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους και δόξα το Θεό, επιτρέψτε μου να πω, μέσα στα πλαίσια ε, της αναφοράς στο Άγιο Πνεύμα που έκανε ο Αντιπρόεδρος, Αλλά αν μπορέσουμε να εκπονήσουμε μεθόδους εκμάθησης γλωσσών, 75 γλωσσών, όχι 25, και 135 που μιλούνται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα διευκολύναμε πάρα πολύ την πρόσβαση. Αν ήταν δωρεάν αυτά τα μαθήματα, ακόμα καλύτερα. Και επιπλέον έτσι θα είχαμε εγγυημένη μια ποιότητα ε, διδασκαλίας παντού για όλους τους φοιτητές κάθε ηλικίας. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα, υπάρχουν πολλά ακόμα και τα πολυμερή έργα συνενώνουν πανεπιστήμια, φορείς, ε, πρωταγωνιστές του κόσμου των γλωσσών και του πολιτισμού και από κοινού εκπονούν προγράμματα και σχέδια για να βελτιώνουν τα συστήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Ποιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί, δεν θα σας διαβάσω τον κατάλογο, αλλά κοιτάξτε, ε, ε, έτσι, θεωρητικά, εντός εισαγωγικών μπορούν οι πάντες να είναι δικαιούχοι. Όχι μόνο τα πολιτιστικά Ινστιτούτα, τα μουσεία, τα μέσα ενημέρωση, τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ ανοιχτέ οι δράσει αυτέ. Παρόλο που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι λιγότερο πολύγλωση από το Κοινοβούλιο, γνωρίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε ε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών για μια σειρά από λόγου, στου οποίου θα επεκταθώ στη συνέχεια αν έχω χρόνο. Πέρα λοιπόν από αυτά τα προγράμματα υπάρχουν και προτεραιότητες. Δηλαδή, αν θέλετε να καταθέσετε μία πρόταση, να υποβάλλετε ένα αίτημα για να επιλεγεί και να χρηματοδοτηθεί θα πρέπει να ανήκει σε κάποια προτεραιότητα. Το ένα έχει να κάνει με τη συνεργασία του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της απασχόλησης, είναι λεγόμενη απασχολησιμότητα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι και μάλιστα θεμελιώδης από πλευράς Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι η προώθηση και ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων σε λιγότερο μιλούμενες γλώσσες που είναι από μικρότερες χώρες, περιφερειακές ε, γλώσσες και ε, μειονοτικές. Ε, τρίτη προτεραιότητα. Γλωσσικές δεξιότητες παντού σε όλο το εύρος ε, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δημιουργία ε, προγραμμάτων, σπουδών, ε, οτιδήποτε μπορεί να διευκολύνει την εκμάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών παντού. Τέταρτη προτεραιότητα, η υποστήριξη στη δίγλωση εκπαίδευση. Είμαστε πεπισμένοι, γιατί έχουν γίνει μελέτες σχετικά, που αποδεικνύουν ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη και χρήσιμη αυτή η δίγλωση εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες από το σχολείο. Είναι αυτό που λέγεται CLIL στα αγγλικά, δηλαδή ε, και το περιεχόμενο και η γλώσσα ολοκληρωμένη. πούμε, δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω, αλλά ε, τη γεωγραφία στα Ιταλικά, ας πούμε, να την κάνουμε στο σχολείο, ή την οικονομία στα Ισπανικά ε, ή στα Αγγλικά. Ε, όταν κάποιος είναι ε, από άλλη μητρική γλώσσα. Αυτά είναι τα προγράμματα λοιπόν τα πολυμερή. Πέμπτη προτεραιότητα, εκμάθηση ε, γλωσσών των γειτονικών χωρών. Γιατί, ότι μπορεί να είναι σημαντικά τα αγγλικά και όλοι να μαθαίνουμε και να μιλάμε αγγλικά, είναι βασική δεξιότητα, που πούμε, δεδομένη όταν κάποιος θέλει να μπει στην αγορά εργασίας ε, των γειτονικών χωρών ή άλλων, έχει σημασία να μιλάει τη γλώσσα του γείτονά του και είναι δύσκολο και περίπλοκο. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να μπορεί να επεκτείνεται και προς την εκμάθηση των γλωσσών των γειτονικών της χωρών. Ερχόμαστε τώρα στα δίκτυα. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Δηλαδή, Έχουμε μια ιδέα έτσι πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, να αυξηθεί και η γνώση και η ποιότητα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι πολλαπλασιαστές για να έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πνεύ που να γίνονται ανταλλαγές πληροφοριών, βελτίστων πρακτικών και να συνεισφέρει αυτή η προσπάθεια στον εξυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Ποιος μπορεί εκεί να συμμετέχει ε, ίσως είναι μικρότερος ο κατάλογος από τις προηγούμενες δράσεις και τα προγράμματα που ε, επικεντρώνονται πιο πολύ στην ουσία και στο περιεχόμενο, αλλά εδώ μπορείτε να δείτε ότι μπορούν να συμμετέχουν πολλοί φορείς και κοινωνική και ε, εκπαιδευτική αλλά και εκτός της παιδείας ε, και φορείς πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης. Όλη αυτή είναι επιλέξιμη. Ποιες είναι τώρα οι προτεραιότητες των δικτύων. Η πρώτη προτεραιότητα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική είναι η ισότητα των ευκαιριών. Η κοινωνική ένταξη συμπραγμανωμένων και των μεταναστών. Είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει κοινωνική ένταξη των μεταναστών να είναι σε θέση να μιλούν τη γλώσσα της χώρας ε, υποδοχής τους αλλά και να μπορούν ταυτόχρονα να ομιλούν και να ε, ασκούν τη ε, μητρική τους γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη αυτός ο πλούτος να μην θεωρείται συνεχώς εμπόδιο, μπορεί να είναι μια επιπλέον δυσκολία, αλλά είναι καλό τελικά και εμπλουτιστικό στοιχείο και απολύτου σημασίας τα κράτη-μέλη να επενδύουν στην απαραίτητη προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για να δημιουργούνται καλύτερες μέθοδοι όσο είναι γυνατό για να ε, γίνεται η διδασκαλία και αυτών των γλωσσών και της χώρας και της περιφέρειας και του τόπου που ζουν οι μετανάστες για να έχουν και δίγλωση εκπαίδευση, όχι μόνο σε ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και στη δική τους. Είναι ο καλύτερος τρόπος ε, συμπεριφοράς απέναντι σε ένα πολίτη σεβασμός. Επόμενη προτεραιότητα, δεύτερη των δικτύων, αυτή είναι λίγο ευρωπαϊκή, πώς να το πω, είναι αμυγός των θεσμικών οργάνων. δεν ξέρω, ε, ένα σήμα ευρωπαϊκών γλωσσών, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, έχει διάφορους χαρακτηρισμούς, είναι αυτά. Αυτά είναι έργα που προέρχονται από τα κράτη-μέλη και εντοπίζουν τα καλύτερα ε, μοντέλα ε, εκμάθησης γλωσσών και τα πολλαπλασιάζουν. Ποια λειτουργούν καλύτερα, ας πούμε. Υπάρχουν σχέδια με πολυγλωσσία ε, η τηλεόραση, η μέσα ενημέρωση, η tv ή δεν ξέρω, στη Γερμανία. Υπάρχουν μια σειρά ε, φορείς και επιχειρήσεις και τομείς στην εκπαίδευση και προσπαθεί κάθε χώρα να εντοπίσει τις καλύτερες αυτές προσπάθειες. Φέτος, σε μια πρόσφατη ε, εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Κύπρο και μας τίμησε με την παρουσία του ο, ο κύριος Μαρτίνης και η κυρία Γενική Διευθύντρια, κυρία Όλγα Κοσμίδου, σε αυτή λοιπόν τη διάσκεψη για πρώτη φορά απονεμήθηκαν τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία σε αυτά τα ευρωπαϊκά σήματα γλωσσών ε, που ε, είχαν προταθεί από τις διάφορες χώρες. Βέβαια αυτό είναι μια δράση εχμής ε, πολύ υψηλής ποιότητας και καταφέραμε την επόμενη φορά να είναι προτεραιότητα λόγω της δυνατότητας του αντικτύπου της ευρωπαϊκής διάστασης και το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα. Αυτά ε, τα προγράμματα προτείνονται από τις εθνικές υπηρεσίες που είναι οι συνομιλητές μας και αμόλογοι για τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Οπότε αν θέλετε να ενημερωθείτε έχετε εδώ ε, τον ιστότοπο ε, για να μπορέσετε αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία. Προτεραιότητα τρίτη. Τα γνωρίζετε. Ε, και από τα προηγούμενα προγράμματα η στήριξη των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, γιατί η στήριξη για τις πολύ μεγάλες παγκόσμιες γλώσσες είναι δεδομένη, είναι γνωστή, είναι συχνή. Αυτό που χρειάζεται είναι να στηρίξουμε τις μικρές γλώσσες μικρών χωρών, τις περιφερειακές και ακόμα και τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Τέταρτη και τελευταία προτεραιότητα των δικτύων που υπάρχει και στα ε, σχέδια τα πολυμερή είναι η δίγλωση εκπαίδευση. Σας είπα ποιο ήταν αυτό και το όνειρό μας θα ήταν να υπάρχει αυτή ε, η εκπαίδευση μέχρι και το πανεπιστήμιο σε όλες τις βαθμίδες από το νηπιαγωγείο, το παιδικό σταθμό, το δημοτικό, το γυμνάσιο και ε, είναι πάρα πολύ όμορφο να είναι κανείς δίγλωσος και πάρα πολύ καλό και το βλέπουμε και από μελέτες ψυχο ε, νευρολογικές και γενικότερα για την ανάπτυξη του ατόμου είναι πολύ ε, καλό να είναι κανείς δίγλωσος. Τώρα, η τελευταία δράση που χρηματοδοτούμε από τις γλώσσες είναι τα συνοδευτικά μέτρα. Τα συνοδευτικά μέτρα, όπως είδαμε, είναι πολύ μικρά ως πρόγραμμα στη χρηματοδότηση. Είναι δράσεις κυρίως ενημερωτικές, πληροφόρησης, επικοινωνίας. Ε, παράδειγμα, πώς μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει διασκέψεις, σεμινάρια, είναι δίκτυα ανταλλαγής καλών πρακτικών, ε, ποιος μπορεί να επωφεληθεί. Ε, η λίστα των δικαιούχων είναι πολύ μεγάλη. Αν έχετε ένα σχέδιο που σας ενδιαφέρει, ε, λίγο να εκθέσετε και να παρουσιάσετε και στους άλλους, μπορεί να χρηματοδοτηθείτε από αυτή τη δράση ή να κάνετε να υποβάλλετε αίτηση υποψηφιότητας. Τώρα, είπαμε τις προτεραιότητες και τα βασικά στοιχεία. Στα ε, πολυμερή προγράμματα είναι η συνειδητοποίηση για τις γλώσσες, βεβαίως η ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων εκμάθησης γλωσσών με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Εδώ όμως δεν εντάσσονται ούτε τα λεξικά ούτε οι βάσεις δεδομένων. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Στα δίκτυα, αυτό που έχει σημασία είναι ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, και η προώθηση ε, της καινοτομίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Στα συνοδευτικά μέτρα, όπως σας είπα, πρόκειται κυρίως για δράσεις ενημέρωσης, επικοινωνίας και πρέπει να γνωρίζετε κάτι πολύ σημαντικό για τις δράσεις αυτές που χρηματοδοτούμε. Ε, όλες οι γλώσσες είναι επιλέξιμες, όλες οι γλώσσες. Έχουμε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εκμάθηση των κινέζικων, τη διδασκαλία των αραβικών, των ρωσικών. Είναι επιλέξιμες όλες οι γλώσσες. Δεν περιορίζεται η δράση αυτή μόνο στις ε, κοινοτικές επίσημες γλώσσες, οι μειονοτικές ή παρούσες, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι επιλέξιμες όλε οι γλώσσε του κόσμου. Τα κριτήρια επιλογής το βλέπετε εδώ, το πόσο υπάρχει σκοπιμότητα, ποιότητα του προγράμματος εργασίας, καινοτομία, η ποιότητα της σύμπραξης κρατών ή του ομίλου πανεπιστημίων ε, που ε, δημιουργείται, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ο λόγος κόστους ωφέλειας, ο αντικτύπος, η ποιότητα διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και η συμμετοχή τρίτων χωρών που έχει σημασία στα μάτια μας. Αν θέλετε λοιπόν να συμμετέχετε σε αυτή τη δράση και να δείτε ό,τι δεν μπόρεσα να σας πω, βλέπετε εδώ τις ιστοσελίδες που θα σας ενημερώσουν και θα βρείτε και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα, προθεσμίες και ό,τι άλλο μπορεί να σας ενδιαφέρει. Πριν σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και αφήσω και πάλι το λόγο στη συντονίστριά μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την πολιτική της πολυγλωσσίας. Να μην περιοριστώ μόνο στη χρηματοδότηση που ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο φυσικά τα χρήματα και η δυνατότητα χρηματοδότησης για τις φιλοδοξίες και τα όνειρά μας, αλλά να πω δύο λόγια για την πολιτική της πολυγλωσσίας, δεδομένου ότι έχουμε την ε, τύχη να έχουμε ενώπιό μας τον ε, αρμόδιο αντιπρόεδρο για την πολυγλωσία που είναι πραγματικά η ενσάρκωση αυτής της πολιτικής. Θέλω να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σήμερα η πολυγλωσία είναι πιο ισχυρή από ποτέ και θα σας το αποδείξω. Για ποιο λόγο. Διότι σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρόσφατα τα τρία θεσμικά όργανα της τριγώνου της κοινοτικής μεθόδου που είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινοβούλιο και Συμβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν να υποστηρίξουν τις γλώσσες ε, στο πιο υψηλό επίπεδο. Οι τρεις λοιπόν που διαπραγματεύονται για τα επόμενα προγράμματα, την επόμενη γενναία προγραμμάτων εκπαίδευσης, ε, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θεωρούν την εκμάθηση γλωσσών και την προστασία της γλωσσικής ποικιλομορφία μία από τις έξι προτεραιότητες του προγράμματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ε, θα αφορά την περίοδο 2014-2020 και ο προϋπολογισμός που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, αν ε, προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, το μέλλον των γλωσσών θα είναι τουλάχιστον καλύτερο από το σημερινό. Αυτό σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για το νέο πρόγραμμα που προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ιδιαίτερα η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου που θεωρεί προτεραιότητα τις γλώσσες. Ε, τα άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο Υπουργών, το Νοέμβριο του 2011 ενέκρινε συμπεράσματα για ε, τις γλωσσικές ικανότητες και την προώθηση της κινητικότητας. Κινητικότητα και για την εκμάθηση γλωσσών αλλά και για εργασία. Αυτό είναι πολιτική εντολή, έτσι το ονομάζουμε με όρους ευρωκρατικούς. Ε, θα πρέπει να δούμε τι συνέχεια δώσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα, εάν υλοποιήσαμε αυτά που μας ζητεί το Συμβούλιο ε, μας καλεί να κάνουμε. Είναι πολιτική εντολή λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου ενέκρινε ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια πάρα πολύ φιλόδοξο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που έρχεται να υποστηρίξει πάρα πολύ τις γλώσσες, όχι μόνο από πλευράς απασχολησιμότητας ή κατάρτισης, αλλά ε, βάζει στο κέντρο τον πολίτη, που άλλωστε αυτό χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία ολόκληρη. Και τέλος, 28 και 29 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λίγο νωρίτερα, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης τόνισαν τη σημασία και την αξία των γλωσσών για την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρώπη. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια κατάσταση ε, για τις γλώσσες. Γιατί συμβαίνει αυτό. Η πολυγλωσία είναι πιο ισχυρή από ποτέ διότι ε, στη διεθνή σκηνή συνεργασία μας με τις χώρες που εμείς ονομάζουμε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κίνα αποφάσισε στη συνεργασία της με την Ένωση να ε, καθορίσει τρεις προτεραιότητες για την ανάπτυξη, για την ε, απασχόληση, γνώμη, που είναι με τη σειρά αυτή οι γλώσσε, η ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση. Συνεργαζόμαστε επίσης με την Ινδία, τη Βραζιλία, ε, την ΑΣΕΜ, Μερκοσούρ και άλλους. Υπάρχει λοιπόν μια διεθνή συνειδητοποίηση της αξία των γλωσσών και είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας. Τώρα, στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη γνωρίζετε ότι πολλές από τις ε, πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη συνέχεια, ε, καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη, όχι όμως ε, στο Συμβούλιο Υπουργών που είναι η επίσημη ε, συνεδρίαση, αλλά σε ομάδες εργασίας, αυτό που ονομάζουμε ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, όπου εκπρόσωποι από διάφορα κράτη-μέλη χαράζουν κοινέ στρατηγικές. Τώρα συστήσαμε μια ομάδα για τις γλώσσες και ό,τι έχει να κάνει με όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στο παρελθόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάτι σχετικό για την απασχολησιμότητα, για τις επιχειρήσεις. Τώρα διανύουμε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ελπίζω και εσείς να μας βοηθήσετε και να μας κάνετε προτάσεις ενδιαφέρουσες που θα μας εκπλήξουν. Τώρα, για τη συνεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Γκράτς και πρόκειται να υπογράψουμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις. Επίσης, ε, έχουμε δύο πλατφόρμες και βλέπω ότι είναι εδώ ο πρόεδρος κύριος Ούβε Μερ της μίας πλατφόρμας και η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις. Γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι η Ευρώπη για να μην είναι μία ε, σκοτεινή γραφειοκρατία θα πρέπει ε, να παραμένει σε στενή επαφή με την κοινωνία και τους ενδιαφερομένους. Κάθε πλατφόρμα απαρτίζεται από εκπροσώπους 30 και πλέον φορέων και μας επισημαίνουν τα λάθη μας, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και πώς μπορούμε να προοδεύσουμε. Ε, και στον επιστημονικό τομέα επίσης, το ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Λόπες, Εκεί έχουμε αυτό τον καιρό μελέτες όπου μπορούν με αξιόπιστα στοιχεία να μας επιτρέψουν να χαράξουμε νέες στρατηγικές και να σχεδιάσουμε νέες στρατηγικές. Ε, Ευρωβαρόμετρο, η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τη Γλωσσομάθεια των Ευρωπαίων και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται ξένες γλώσσες στα ευρωπαϊκά σχολεία. Τώρα, πάρα πολύ πρόθεσμα. ποιες είναι οι προτεραιότητες της πολιτικής πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο για το δικό μου θεσμικό όργανο μιλώ. Δεν θα τολμούσα ποτέ να το κάνω για άλλο θεσμικό. Τις επόμενες μέρες θα εγκριθεί μια πολύ φιλόδοξη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τίτλο «Αναθεωρώντας την εκπαίδευση». είναι έγγραφο εργασία των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τι γλώσσε. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η διοργάνωση μια διάσκεψης που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική και για εσά πιστεύουμε και θα ήθελα να σα καλέσω να συμμετέχετε στο Πεκίνο την 1η Δεκεμβρίου, είναι ημέρα Σάββατο. Και οι φίλοι μα οι ε, Κινέζοι εργάζονται όλο το Σαββατοκυριακό, θα του ακολουθήσουμε και εμεί αυτό το δρόμο. Την 1η Δεκεμβρίου λοιπόν με στόχο να οικοδομήσουμε μια συνεργασία με τους φίλους μας στην Κίνα για να μπορέσουν σε ένα πρώτο στάδιο να έρθουν στην Ευρώπη να μάθουν τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες που στη δική τους ε, αντίληψη και ορισμό είναι όλες οι γλώσσες πλην των Αγγλικών. Επίσης να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας. Η οικογένεια των γλωσσών είναι οι γλωσσικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μετάφραση και διερμηνία, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές είναι λοιπόν οι προτεραιότητές μας και ελπίσουμε όλα να πάνε όπως τα σχεδιάσαμε. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με βεβαίως στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση τυχόν έχετε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας κυρίως. Teşekkür e, Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Ιζαμπέλα Μπατιού που εδώ και χρόνια είναι υπεύθυνη για τις ε, του, του τμήματος Ερμηνείας του Πανεπιστημίου της, του Κλούζ και είναι σήμερα επικεφαλής της Ρουμανικής, ε, μετάρχης της Ρουμανικής ε, Διερμηνίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά είναι για μένα να μπορώ να μιλήσω σήμερα στα ρουμανικά και κυρίως για να μεταφράσω σε πραγματικότητα την αρχή που μας ε, συγκεντρώνει όλο σήμερα εδώ, δηλαδή την πολυγλωσία. Για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αυτή η αρχή πολύ συχνά ε, την επικαλούμαστε ως κάτι το αφηρημένο, ξεχνώντας ε, πόσο είναι απτή η αρχή αυτή, το να μιλήσουμε στην ίδια μας τη μητρική γλώσσα, να εκφράσουμε δηλαδή ε, τα βαθύτερα νοήματα, είναι μια χειρονομία, ένα άνοιγμα προς τους άλλους και για μένα σήμερα, γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη τιμή που μπορώ να απευθύνομαι σε ένα τόσο διακεκριμένο κοινό στη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να πω ότι εγώ μιλώ μια γλώσσα η οποία δεν είναι πολύ διαδεδομένη, αν και η Ρουμανία είναι μια χώρα μεσαίου μεγέθου, σύμφωνα με τι στατιστικέ. Έχει γίνει επίσημη γλώσσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 2007 και έπειτα σε προσωπικό επίπεδο ω υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω δει είναι, πόσο περίπλοκο είναι ο χαρακτήρα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόσφατό μου παρελθόν ωστόσο παραμένει συνδεδεμένο με τον ακαδημαϊκό κόσμο, γι' αυτό και έχω μια διπλή ευαισθησία. Ε, διπλή ευαισθησία ω ερμηνέα και ω ακαδημαϊκός και γι' αυτό και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα όσα είπαν οι διάφοροι συνάδελφοι, επιστήνοντα την προσοχή σα σε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που ε, ανοίγει στον ακαδημαϊκό κόσμο η διερμηνία συνεδρίων. Δεν έχω και πολλά να πω γιατί έχουν μιλήσει οι ήδη. Είναι σαφές ότι το Εράσμος Μούντους, ο ξάδερφος του Εράσμους, έχει τη δυνατότητα να ε, φέρει σε επαφή τα πανεπιστημιακά περιβάλλοντα συμφωνούμε όλοι και πρόσφατα ο τύπος το έχει συστηρίξει αυτό και λέει πως τα προγράμματα αυτά είναι επιτυχή γιατί επί τη βάση αυτό και υπάρχουν στατιστικές έχουν δε παρουσιαστική κάποια στοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν πως η πολυγλωσία είναι ζωντανή και μεταφράζεται στην καθημερινή ζωή ε, χιλιάδων φοιτητών. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα Εράσμος και αυτοί οι φοιτητές, οι τότε φοιτητές είναι πια επαγγελματίες εργαζόμενοι. Στις αρχές του έτους ο Ουμπέρτο Έκο είπε το εξής, ότι το Εράσμος δημιούργησε την πρώτη γενεά των πραγματικών γνήσεων Ευρωπαίων νέων. Και ακόμα και αν ακούγονται που και που φωνέ που λένε πω το πρόγραμμα Εράσμο χρησιμοποιείται περισσότερο για τουρισμό και όχι για μελέτη, όσοι παρακολουθήσαμε την ανάπτυξη του προγράμματο, την εξέλιξή του και έχουμε συντονίσει το πρόγραμμα αυτό στα διάφορα πανεπιστήμια μα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το να ζούμε αλλού και να σπουδάζουμε αλλού δεν είναι κάτι το αντιφατικό. Ίσα ίσα μόνο με μία ε, βήθηση στη γλώσσα, με μια βαθιά βουτιά, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί πλήρως το γεγονός ότι βρίσκεται στην ε, χώρα. Και αυτό αποδεικνύεται και από τους ε, φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το Εράσμους. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σημαντική η γνώση των ξένων γλωσσών και όσοι την είχαν, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα Εράσμους δείχνουν και αυτό το είδος την ευελιξία, την κινητικότητα Αυτά τα στοιχεία μπορεί να σας να φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά επιστημονικά, αλλά σας εγγυώμαι ότι αυτά στηρίζονται από συγκεκριμένες έρευνες και ότι η φοιτητική κινητικότητα έχει αποτελέσει πλέον, μάλλον αποτελεί πλέον ένα θέμα ακαδημαϊκής έρευνας, όπως η οικονομία, οι διάφορες επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως η κινητικότητα είναι εξάλλου ένα, μια προϋπόθεση για το επάγγελμα του διερμηνέα. Πώς μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε στους ε, νέους φοιτητές που θέλουν να γίνουν διερμηνείς τη δυνατότητα να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, πέρα δηλαδή από τις δυνατότητες που τους προσφέρουν αυτά τα προγράμματα. Και μάλιστα το ίδιο τα πανεπιστήμια θα πρέπει να τους προωθήσουν, ε, στηρίζοντας ε, προγράμματα σπουδών όπως τα μεταπτυχιακά για τη διερμηνία. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι οι εξελίξεις μπορούν να είναι πολλαπλές και θα σας δώσω τρεις ε, άξονες από τη μεγάλη γάμα δυνατοτήτων που ανέφερε η κυρία Μπελέντη Κυρός για παράδειγμα, όσον αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο και τη σύνδεσή του με τα πανεπιστήμια. Δεν αφορά αυτό μόνο μαθήματα ξένων γλωσσών, αλλά και μαθήματα δερμηνίας, μετάφρασης καλής ποιότητας για τα πράγματα για τα οποία χρειάζονται επαγγελματίες με συγκεκριμένες δεξιότητες. Έπειτα για τις λιγότερο διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες, τις περιφερειακές γλώσσες, χρειάζεται μια γλωσσική και πολιτιστική διαμεσολάβηση ανάμεσα σε μια μειοψηφία και μια πλειοψηφία. Και αυτό είναι μέρος της δουλειάς του διερμηνέα. Τέλος, τα δίκτυα που δίνουν ε, ζωή στις ε, γλωσσικές πολιτικές. Το θέμα δηλαδή την έννοια του networking, της δικτύωσης και είναι αυτό ένα σημαντικό στοιχείο της διάσκεψής μας από όλα τα διάφορα μαθήματα που αφορούν ε, πολυμερή μάθηση γλωσσών, ε, μεταπτυχιακά και σπουδές, ε, δυνατότητες διάδρασης και αλληλεπίδρασης. Εγώ να μιλήσω το, το, για το ευρωπαϊκό πτυχίο, μεταπτυχιακό, στο, στη Διερμηνία. Βασίζεται στην εγγύηση της ποιότητας ως κριτήριο Πρόκειται για μια ευέλικτη μορφή πανεπιστημίου, ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, ε, καλή και παροτρύνει στην επιστημονική έρευνα και προσφέρει επίσης στους φοιτητές ένα διπλό δίπλωμα. Θα είχαμε πολλά ακόμα να πούμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διάφορα πτυχία που προσφέρονται. Δεν έχω όμως το χρόνο και γι' αυτό θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δεύτερη πιο αγαπημένη μου γλώσσα που είναι η γαλλική θα ήθελα να σας ε, προτείνω μια ε, άσκηση, να σημειώσετε ένα σύντομο κατάλογο λέξεων κλειδιών και σας τις αναφέρω. Διεθνοποίηση, όμιλος, ετικέτα, κινητικότητα, δίκτυο, εταιρικότητα, αριστεία, ελκυστικότητα, ανταγωνιστικότητα, εξασφάλιση, σύγκληση και καλές πρακτικές. Τώρα διοργανώστε τις αυτές σε συγκεκριμένα νοήματα. Μετρήστε την έννοια, τις έννοιες αυτές μέσα στην οικονομία του δικού σας, δικού τμήματος και δείτε πώς αυτές σχετίζονται με το μέλλον των φοιτητών σας. Δείτε, ας πούμε, κάντε ένα peer review. Ποσοστοποιήστε και η χρήση των στατιστικών. Εδώ είναι ε, ε, απαραίτητη. Ελάτε σε επαφή με τους ε, συναδέλφους σας και συγκρίνετε αυτές τις ε, έννοιες. Ενδεχομένω ξανακάντε την ίδια προσπάθεια και χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όπως ε, η μεταπτυχιακή στο διερμηνία συνεδρίων στο δικό σας τμήμα. Και έπειτα να μην ξεχάσετε να συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία των συναδέλφων σας στην τρίτη σύνοδο των Πριτάνεων για να δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα çok teşekkür ediyorum. Σε ευχαριστούμε, Ιζαμπέλα. Όντως, το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και σίγουρα το οικονομικό τμήμα είναι πολύ σημαντικό επίσης για προγράμματα όπως ε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο και έχουμε συμπεριλάβει και νέους τομείς ε, στα δίκτυα αυτά και για όλα τα δίκτυα φυσικά η χρηματοοικονομική πτυχή έχει θεμελιώδη σημασία γι' αυτό και ήταν απαραίτητο να την εξετάσουμε και σήμερα. Και για πολλές χώρες ε, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι πολύ κέριο ζήτημα. Υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ. Λοθάνο, de la Ραφαέλο Σάνα από το Πανεπιστήμιο τη Μπολόνια στην Ιταλία. Eh, Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα που ανακύπτει σε τέτοιου είδους ε, συναντήσεις. Αφενός μιλούμε για πολυγλωσία, ακούμε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα και μάλιστα με το βλέμμα μας στραμμένο προς το μέλλον, αλλά ας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώ εννοώ. Πριν από ένα-δύο χρόνια, δεν κάνω λάθο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων την εκπόνηση μια μελέτη για την ε, πολυγλωσία. Ένα από τα βασικά πορίσματα τη μελέτη ήταν ότι ο ε, κάθε Ευρωπαίο πολίτη θα πρέπει πέραν τη μετρική του γλώσσα να γνωρίζει τουλάχιστον δύο ακόμη γλώσσε. Και μάλιστα έλεγε να υιοθετήσει μία γλώσσα μειονότητα και κάτι τέτοιο. Περίπτωση της Ιταλίας. Την ίδια χρονιά που δημοσιεύθηκε η έκθεση αυτή, γίνεται μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, όπου εισάγει την ε, ενιαία γλώσσα, μία μόνο γλώσσα για όλη την παιδεία, τα εγγλικά. Η κυρία Δεκαιρός μίλησε για την κατάσταση αυτή ε, και την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την πολυγλωσσία. Αλλά σε επίπεδο πανεπιστημιακό το θέμα της πολυγλωσσίας είναι ένα ζήτημα που έχει ενταχθεί αρκετά και αποτελεί κάτι πολύ κοινό γιατί όλα, απ' την άλλη βέβαια όλα τα πανεπιστήμια έχουν μαθήματα και μεταπτυχιακά στα αγγλικά σχεδόν αποκλειστικά σαν να μην υπήρχαν οι άλλες γλώσσες. Υπάρχει λοιπόν όπως βλέπετε μια διαφοροποίηση μεταξύ της προετοιμασίας του απλού πολίτη, προκειμένου να ε, ή του νέου, νέου πολίτη προκειμένου να ανελιχθεί και να ε, ενηλικιωθεί και να σπουδάσει και να ε, σπουδάσει και στο πανεπιστήμιο και τις έλλειψη στο μέσο που υπάρχουν μερικές φορές για κάτι τέτοιο. Ναι, όντως, είναι αυτό που στην κοινοτική ορολογία αποκαλούμε στόχο της Βαρκελόνης όπως προσδιορίσε το Συμβούλιο του Μαρτίου του 2002 στη Βαρκελονική, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρότειναν να βοηθήσουν κάθε Ευρωπαίο πολίτη για να μάθει δύο ξένες γλώσσες πέραν της μητρικής του γλώσσας. Η κατάσταση στην Ιταλία είναι αυτή που μας περιγράψατε. Βέβαια το θέμα της γλωσσικής πολιτικής και στην παιδεία και στην κατάρτιση και επιμόρφωση είναι εθνική αρμοδιότητα. Η, κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Εμείς ε, ε, ενισχύουμε ίσως τις προσπάθειες των κρατών μελών, συνδράμουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προβλέψουμε στόχους ε, της πολιτικής της παιδείας ή της πολιτικής και της γλώσσας στην, ε, στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί κανείς να μάθει 54 διαφορετικές γλώσσες. Δεν έχει επιλογή μία κύρια γλώσσα. Στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Βραζιλία για παράδειγμα, αποφάσισαν με νόμο του 2005 ότι η πρώτη ξένη γλώσσα στα σχολεία θα είναι τα ισπανικά. Γιατί είναι μια χώρα που έχει επίσημη την Πορτογαλική σε, σε μια ήπειρο που μιλάει εξοχήν τα ισπανικά. Οπότε ε, τελικά, επειδή και τα αγγλικά έχουν μεγάλη παρουσία, ουσιαστικά βγαίνουν οι φοιτητέ μιλώντα τρει γλώσσε. Αλλά ω προ αυτό που είπατε, έχετε πραγματικά δίκιο. Μία ακόμη ερώτηση θα ακούσουμε και μετά θα ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όντω ε, υποστηρίζει κάποια μαθήματα στα αγγλικά, θα πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ιδεαλιστέ αλλά και ρεαλιστέ. Δηλαδή, αυτό που λαμβάνουμε στο Erasmus Mundus, το 85% των projects είναι στα αγγλικά. Και δεν είναι αυτό κριτήριο επιλεξιμότητα. Τα πανεπιστήμια γνωρίζουν ότι αν θέλουν να προσελκύσουν φοιτητέ από την Κίνα, την Ινδία ή την Ιαπωνία, δεν έχουν άλλη δυνατότητα παρά να προσφέρουν μαθήματα στα αγγλικά. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να προωθήσουμε και άλλες ε, ευρωπαϊκές γλώσσες, μέσω του πολιτισμού, μέσω κάποιων μαθημάτων, όπως είπαμε και στα πλαίσια του Erasmus Mundus, να ε, θέσουμε ως υποχρεωτική την εκμάθηση και άλλης γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών, πέραν των αγγλικών δηλαδή. Η Όλγα. Όργα Γκρεγόρβα από την Ρωσία, από Πανεπιστήμιο τη Ρωσία. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Τεγκερός και την ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα παρουσία της. Για ποια από τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να ήταν επιλέξιμη και η Ρωσία. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε την ερώτησή σας στα ρωσικά. Θα μπορούσατε κάλλιστα να διατυπώσετε την ερώτησή σας στα ρωσικά. Πολύ ευχαρίστω, γιατί έχουμε και διερμηνία από τα ρωσικά. Α, θέλετε να επαναλάβω την ερώτησή μου στα ρωσικά. Μάλιστα. Ονομάζομαι Όλγα Γκρεγόροβα από το Πανεπιστήμιο του Αστραχάν στη Ρωσία. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Τικεϊρός που μας έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Μα παρουσιάσετε μια πληθώρα προγραμμάτων. Σε ποια από αυτά θα μπορούσε να συμμετέχει και η Ρωσία. Σε όλα. Σε όλα. Έχω πολύ καλά μαντάτα. Η Ρωσία είναι επιλέξιμη για όλα τα προγράμματα. Και αν δεν κάνω λάθος υπάρχει ένα πολύ καλό α, σχέδιο συνεργασίας α, υπό την αιγύδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ ε, Κωνσταντινούπολη, Σταμπούλ και Αστραχάν. Σα εθαρρύνουμε λοιπόν να συνεχίσετε ε, και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος, πιο ευχάριστη νότα για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ, αν και μας έμεινε χρόνος για μία ακόμη ερώτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα κροατικά. Είμαι από το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπ και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχω αυτή την ευκαιρία σε αυτή την ομίγυρη να χρησιμοποιήσω τη μετρική μου γλώσσα. Δεν νομίζω ότι η προστασία της ε, πολυγλωσσίας είναι αντιφατική με την ε, ύπαρξη και μιας Λίγκου φράγκα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ανέκαθεν υπήρχε κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι το 90% της ε, αλληλογραφίας είναι διμερής και χρειαζόμαστε μια τέτοια κοινή γλώσσα, Λίγκου φράγκα, στη πιο βασική της μορφή. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ έχει αποφεληθεί πολύ από το πρόγραμμα της ε, πολυγλωσίας, γιατί χάρη σε αυτό διοργανώσαμε το μεταπτυχιακό μας ε, στην, ε, για τη διερμηνία στο Ζάγκρεπ. Και έτσι κάναμε την επιμόρφωση των διερμηνέων μας, που αλλιώς δεν θα είχαν την ευκαιρία να εργαστούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο διερμηνίας, σπουδών διερμηνίας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα τέτοιο δίκτυο για σπουδές διερμηνίας. Μήπως θα μπορούσαμε μια τέτοια πρόταση να την προωθήσουμε. Κύριε Μαρτίνεφ, δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθό τώρα να παρέμβω εγώ στη συζήτηση, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο φίλος μας από την Κροατία. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και με ανησυχεί αυτό το ζήτημα της lingua franca. Πρώτον, τι θα πει lingua franca. Είναι μια γλώσσα για να μπορεί κανείς να επικοινωνεί με το σύνολο των πολιτών. Μα ήδη έχουμε αποδείξει αρκετά ότι το 90% παγκοσμίως, ας πούμε, ε, ε, θα ήταν 999 της χιλής των πολιτών που θα έμεναν στο περιθώριο της περίφημης ε, lingua franca. Και επίσης κάτι άλλο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το θέμα δεν είναι lingua franca, είναι lingua unica και η ενιαία γλώσσα είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Φορέας αυτό που ονομάζεται ενιαία σκέψη και ενιαία και μοναδική σκέψη είναι εξορισμού μια σκέψη και ένας φορέας ολοκληρωτικής δράσης στις κοινωνίες μας. Και επειδή εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι προς η αδίποτε ολοκληρωτική σκέψη, γιατί η φύση μας είναι βαθιά δημοκρατική, δεν πιστεύουμε καθόλου στην ενιαία η μοναδική γλώσσα και έχουμε πολλές επιφυλάξεις σε σχέση με την ίδια την έννοια της lingua franca. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. ενδεχομένω να είναι προσωπική ε, άποψη με την οποία συμφωνούν πολλοί συνάδελφοί μου. Αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και τον προβληματισμό. Μήπως lingua franca, ίσον lingua unica και ενία και μοναδική σκέψη είναι μονα... κάτι που οδηγεί σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και κόσμο τελείως διαφορετικό και τελείως αντίθετο από αυτό που έχουμε ε, προσιλωμένοι εμείς ε, την πάλη και τον αγώνα μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με ολοκληρωτικό τρόπο τώρα θα κηρύξουμε το πέρας ε, της ενότητας αυτής, γιατί θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη. Сергей Гончаров, э, университет. Э, Сергей Λαγκοντσάροφ από το Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Θα ήθελα να επισήσω την προσοχή των συναδελφών σε ένα από τα ζητήματα κλειδιά που μας απασχόλησαν σήμερα για το θέμα της γλωσσικής ποικιλία και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Λόπες και νομίζω μπορούμε να το συνεχίσουμε και στην επόμενη ενότητα. Ε, έχει σημασία πιστεύω να επικεντρωθούμε ακριβώς σε αυτό το τομέα. Όταν γίνεται λόγος για πολυγλωσία υπάρχουν πολλές πτυχές. Στο πανεπιστήμιο όμως μπορεί κανείς να σπουδάσει ε, ε, να μάθει 40 γλώσσες και οι περισσότερες, οι μισές ε, και πλέον, είναι γλώσσες που μιλούνται από μειονότητες. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα που θα πρέπει να ενισχύσουμε, να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε ε, προς αυτή την κατεύθυνση και αξίζει τέτοια προγράμματα να υποστηρίζονται για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων πολιτισμών. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για καλύτερο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό ε, το θέμα εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες σε τούτο το πάνελ και προχωρούμε αμέσως στην επόμενη ενότητα. vielen herzlichen Dank an... Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη ε, του πάνελ και την Εμπρούντιρικε πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε στο δείπνο, το οποίο δεν αρχίζει αμέσω όμω. Βερνούμε στην επόμενη ενότητα, υπηρεσίε, διερμηνίας και πανεπιστήμια, μια εταιρική σχέση για το μέλλον. Παρακαλώ ε, τα μέλη του πάνελ που δεν είναι ακόμα στο Προεδρείο να έρθουν την Πατρίσια Ρίζου από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κλέρ Ντόνοβαν του ΟΣΑ και τη Σάλι Μπέιλι από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Άλισον Γκρέιβ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Good afternoon. Is everyone awake? Καλησπέρα σας. Είστε όλοι ξύπνοι, δεν έχουμε άλλο διάλειμμα για καφέ. Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Βγαίνει και ο ήλιος, πολύ καλό σημάδι αυτό. Και το πρώτο που μου είπαν να κάνω είναι να δώσω το λόγο στην κυρία Όλγα Κοσμίδου και με πολύ μεγάλη χαρά το πράττω. Παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Είναι περιττό να σας πω πώς είναι η χαρά μου που σας βλέπω όλους σήμερα εδώ. Όχι μόνο γιατί με τους περισσότερους από εσά είμαστε πια μετά από τόσα χρόνια, πολύ παραπάνω από συνάδελφοι, είμαστε φίλοι. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας λόγος. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την οργάνωση του συνεδρίου. Οι συνεργάτες μου και εγώ σκεφτήκαμε πάρα πολύ ως προς τη μορφή που θα έπρεπε να είχε. Διότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να επαναλάβουμε κάτι που οι συνάδελφοί μας της Κομισιόν κάνουν ήδη πολύ καλά. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο οι συνάδελφοί μας της Κομισιόν οργανώνουν μία, ε, μία συνεδρίαση με τα πανεπιστήμια. Αυτό που οργανώσαμε σήμερα είναι κάτι που από όσο γνωρίζω, και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά για την διερμηνία, από όσο γνωρίζω είναι μοναδικό στο είδος του. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν η ιδέα μας ήταν να συγκεντρώσουμε όλους τους πρωταγωνιστές στη δύσκολη υπόθεση της διερμηνίας. Να φέρουμε μαζί τους επαγγελματίες επικεφαλής των μεταφραστικών τμήματων με τα πανεπιστήμια και εν γέννη με τον κόσμο των γλωσσών στην αρχή λοιπόν είχαμε σκεφτεί να έχει αυτή τη μορφή πανεπιστήμια συν οι συνάδελφοι επικεφαλής διερμηνίας και μετάφρασης. Σκεφτήκαμε όμως μετά ότι η εκπαίδευση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να βρούμε διερμηνείς σε όλες τις γλώσσες οφείλεται στο γεγονός ότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση του θέματος της διερμηνίας και της μετάφρασης ότι είναι τομείς στους οποίους χρειάζεται να εκπαιδευτεί κανείς ειδικά και ότι δεν αρκεί να έχει κανείς ένα πτυχίο γλωσσών, ε, λογοτεχνίας ή φιλολογίας μιας γλώσσας, για να μπορεί να είναι καλός μεταφραστής ή καλός διερμηνέας. Αυτό σήμαινε λοιπόν ότι έπρεπε να ευαισθητοποιήσουμε και τους εκπροσώπους των κρατών. Και βεβαίως επειδή δεν είναι πολύ απλό να φωνάξουμε τους υπουργούς, καλέσαμε εδώ και τις μόνιμες αντιπροσωπείες. Αυτό λοιπόν που βλέπετε σήμερα εδώ είναι εκπρόσωποι των κρατών, των κρατών μελών, των υποψηφίων χωρών και των χωρών των οποίων η γλώσσα χρειάζεται στη διεθνή διπλωματία, όπως είναι τα αραβικά, τα ρωσικά, τα κινέζικα, εκτός λοιπόν από τις γλώσσες των υποψηφίων χωρών. Είναι λοιπόν μια μορφή που όπως λέω δεν έχει προϋπάρξει ποτέ. Να συγκεντρώσουμε όλους τους μεγάλους συμμετέχοντες στην υπόθεση της γλωσσικής προετοιμασίας, ούτω ώστε η μετάφραση και η διερμηνία να αναγνωριστούν σε όλα τα κράτη σαν τομείς εκπαίδευσης ξεχωριστά από οποιονδήποτε άλλο, αλλά στο επίπεδο που τους αρμόζει. Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε όθηση σε όλους αυτούς που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε σε καλά ελληνικά major players ε, ή αν θέλετε ε, όλους αυτούς που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, να τους δώσουμε μία όθηση για να συνεργαστούν. Δεν έχουμε την αντίποση ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με μία συνάντηση. Ξέρουμε όμως ότι όλοι όσοι είναι εδώ είναι πεπισμένοι για την αξία αυτού του εγχειρήματος και έχουν οι ίδιοι μεγάλες δυνατότητες ο καθένας στον τομέα τους. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι η σημερινή και η αυριανή συνεδρίαση δεν θα βασιστεί μόνον σε ομιλίες. Όσο καλές και αν είναι αυτές, όλοι σας είστε εξπέρ σε αυτό που κάνετε και δεν νομίζω ότι θα μάθετε πάρα πολλά. Αυτό που ελπίζουμε είναι να δώσουμε μία όθηση στη δικτύωση, στο networking, σε όλα τα σχετικά θέματα. Και αυτό που προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε στο πρόγραμμά μας είναι μία ποικιλία μεταξύ του, της εγρήγορσης, της εκπαίδευσης, της χρηματοδότησης, ήταν το θέμα που είχαμε προηγουμένως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπου και εκεί χρειάζεται δικτύωση. Αύριο, όπως θα δείτε στο πρόγραμμα, θα έχουμε ειδικού έξω από το δικό μας χώρο που θα μας μιλήσουν για το τι συμβαίνει στο μυαλό ενός διερμηνέα όταν διερμηνεύει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε όλοι μας τι μας συμβαίνει όταν διερμηνεύουμε. Θα έχουμε καθηγητές οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τις νέες τεχνολογίες, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, οι νέες τεχνολογίες είναι κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον του επαγγέλματος. Όχι διότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αντικαταστήσουν στο άμεσο ή στο προβλεπόμενο μέλλον τους επαγγελματίες, μεταφραστές ή διερμηνείς, αλλά πρώτον, διότι είναι σημαντικό να καθορίσουμε μόνοι μας τα πλαίσια που χρειάζονται για την συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και να μην το κάνουν άλλοι για μας. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι έχει να μας προτείνει η επιστήμη, να ξέρουμε τι μπορούμε να δεχθούμε και τι όχι. Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την τεχνολογία και βεβαίως δεν είμαστε εμείς που θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και γι' αυτό θα θέλαμε και τα πανεπιστήμια να δώσουν έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις, δεδομένου ότι οι νέες γενιές γεννιούνται και στην κούνια τους έχουν ένα iPhone. Εκεί που σε εμά μας δίνανε μία πιπίλα και μία κουδουνίστρα, στα μωρά τους δίνουν ένα iPhone και βλέπετε ότι μόλις μπορούν να κάνουν ορισμένες κινήσεις και τους δώσετε ένα iPhone, ήδη προσπαθούν να μεγαλώσουν την εικόνα. Είναι κάτι το οποίο με εξέπληξε όταν είδα την κόρη μιας φίλης μου η οποία είναι 11-12 μηνών άρπαξε το iPhone μου και προσπαθούσε να μεγαλώσει την εικόνα. Και κατάλαβα τότε ότι αυτά που η δικιά μας γενιά θεωρεί δύσκολα ή αδύνατα, σε λίγο καιρό θα υπάρξει ένα καινούριο κενό μεταξύ της δικιάς μας γενιάς ή ακόμη και των σημερινών νέων και αυτών που είναι σήμερα μωρά όλους λοιπόν αυτούς τους τομείς θέλησα να, τους να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύνθεση μεταξύ επαγγελματιών που ξέρουν ακριβώς τη δουλειά τους. Ξέρουν ποια είναι τα πλαίσια, ξέρουν ποια είναι τα ζητούμενα και ξέρουν κυρίως ότι δεν θέλουν άλλοι να τους υπαγορεύσουν τι θα είναι η δουλειά τους, πώς θα είναι η δουλειά τους και πώς θα είναι το μέλλον τους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο γιατί δουλεύουμε καθημερινά εδώ και λίγο καιρό σε 24 γλώσσες, για να μην πω σε 25-26 δεδομένου ότι βάσει των στατιστικών μας, πέρσι δεν υπήρξε εβδομάδα στην οποία να μην έχουμε ρώσικα κάθε δύο σχεδόν εβδομάδες είχαμε αραβικά και πολύ συχνά είχαμε κινέζικα. Όχι λοιπόν μόνον γιατί εργαζόμαστε καθημερινά σε τόσες γλώσσες, αλλά διότι έχουμε διαφόρων ειδών εμπειρίες. Είδατε προηγουμένως ότι καθόταν εδώ η κυρία Μπαντιού, η οποία ήταν υπεύθυνη για εκπαίδευση διερμηνέων στο Κλούς και τώρα είναι προϊσταμένη του Τμήματος Ρουμανικής Διερμηνίας στο Κοινοβούλιο. Θα ακούσετε αύριο την κυρία Δάρα να σας μιλάει για θέματα τεχνολογιών. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυνατότητα η οποία μας αναγνωρίζεται από αυτούς που είναι το πιο σημαντικό για μας να αναγνωρίζεται. Βεβαίως από τις αρχές μας, αλλά κυρίως από τους συναδέλφους μας. Και έχουμε επισκέψεις, αναφέρθηκαν προηγουμένως στο Ινδικό Κοινοβούλιο, είχαμε επανειλημμένες επισκέψεις εδώ από το Ινδικό Κοινοβούλιο που μας ζήτησε βοήθεια για να οργανώσει τις εργασίες του με βάση αυτά που γίνονται εδώ και η γενική μου διεύθυνση είχε την τιμή να στείλει επανειλημμένος εκπροσώπους της στο ΠΑΠ, που δεν είναι ο Πάπας αλλά είναι το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στη Νότιο Αφρική, για να τους βοηθήσουμε επίσης να οργανώσουν τη διερμηνία σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν δεν κάνω λάθος η κυρία Πίτ θα μας πει ότι το ίδιο έγινε νομίζω και με θέματα μετάφρασης ε, όχι μόνο με θέματα διερμηνίας. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη τεχνογνωσία στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Αυτή η τεχνογνωσία θα ήταν πολύ στενόμυελο, βρίσκω, να περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση της καθημερινής μας εργασίας. Τα γλωσσικά επαγγέλματα και ιδιαίτερα η διερμηνία είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν περιορίζεται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αν μη τι άλλο, διότι όλοι μας χρησιμοποιούμε λίγο πολύ τους ίδιους φριλάνς διερμηνείς. Ένα φυλά διερμηνέα μπορεί να δουλεύει αυτή τη βδομάδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την άλλη εβδομάδα για το Συμβούλιο τη Ευρώπη, την επόμενη εβδομάδα ε, για το Άρτε ή για το, στο Μόναχο για το πατέντ, ε, για τον οργανισμό ε, ε, που δίνει την certification ή για τα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη ή στη Νέα Υόρκη. Είναι λοιπόν ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορείς να του βάλεις στενά σύνορα στο πλαίσιο μιας και μόνο οργάνωσης. Και ναι, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν αρκετοί καλοί διερμηνείς για να εξυπηρετήσουν όλες τις οργανώσεις, ιδίως αυτές που χρειάζονται τις ίδιες γλώσσες ή αυτές που είναι κοινέ γλώσσε μεταξύ όλων των οργανισμών. Μια ζωή λοιπόν τραβούσε ο καθένα την κουβέρτα προς τη δικιά του τη μεριά. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι έτσι δεν προχωράμε. Αντίθετα πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντες. Είμαι πολύ ευτυχής που είναι εδώ σήμερα, εκτός από όλους όσους ανέφερα, και η ΑΕΚ η πρόεδρος της ΑΕΚ, που έχουν τεράστια εμπειρία σε θέματα αυτά, καθώς και εκπρόσωποι του προσωπικού της Δελεγκασιών των Μονίμων Διερμηνέων και εκπρόσωποι της Επιτροπής Προσωπικού για να δουν μαζί μας ότι θέλουμε να διευρύνουμε τους οριζοντές μας και αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε είναι περισσότερη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες διερμηνίας που το επιθυμούν και τις σχολές. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στο οποίο αντί να κάνουμε όπως γινόταν μέχρι σήμερα που κάνουμε αν θέλετε, εκπαίδευση διερμηνέων μέσω video conference, δηλαδή συνδέεται το κοινοβούλιο με δύο ή τρεις σχολές για να κάνει την εκτίμηση της δουλειάς των φοιτητών. Αυτό που θα προτείνουμε σήμερα είναι να συνδέεται το κοινοβούλιο με μία ή δύο σχολές και έναν άλλο διεθνή οργανισμό και να γίνεται η αποτίμηση ταυτόχρονα από δύο διεθνείς οργανισμούς. Βεβαίως, αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί όπως είπα είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα χάρη στο γεγονός ότι έχουμε την πολιτική υποστήριξη από, τους, τα πολιτικά όργανα και για τα οποία και τους ευχαριστούμε. Νομίζω ότι όλοι μας είτε είμαστε στο μετερίζει της διδασκαλίας της διερμηνίας, είτε είμαστε στο μετερίζει του service provider. Έχουμε τις ίδιες αγωνίες και τους ίδιους στόχους. Και σε ένα επάγγελμα, το οποίο, όπως είπα, είναι ένα επάγγελμα παγκόσμιο, global, οι απαντήσεις δεν μπορούν παρά να είναι συνολικές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ήταν αυτή η συνάντηση πρώτη στο είδος της και σας ευχαριστώ όλους που με την παρουσία σας εδώ την καταστήσατε δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Σε ευχαριστούμε θερμά, Όλγα. Ε, μας ε, περιέγραψες πολύ όμορφα αυτό το πάνελ που ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ ζωντανό και διαδραστικό γιατί κατά την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης είχαμε ε, σκεφτεί να αφήσουμε αρκετό χρόνο σε όλους ώστε να ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους και αυτό είχε κατά νου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, μας προσκάλεσε σε αυτή την άνευ προηγουμένου διοργάνωση με τόση ευγένεια. Καλό θα ήταν να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας σύντομα και μετά να έχουμε μία ζωηρή ανταλλαγή απόψεων, ε, ερωταπαντήσεων. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Ε, συνεχίζοντας το πάθος που έδειξε προηγουμένως ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες και θα μιλήσουμε, όπως είπε και ο Στεφάν Λοπές, για το έργο της ε, γεφύρωσης των πολιτισμών. Αυτό είναι το έργο του Διερμηνέων. Ο Έρμαν Μπόρμπεκ, ένας Αμερικανός συγγραφέας, ε, μίλησε ε, για την σπιτονικοκυρά με πολύ χιούμορ και αναγάγοντάς την σε θεά της αιστείας. Είπε η μητρότητα το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο φυσικά αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Το τρίτο ήταν η διερμηνία, το τέταρτο ήταν ε, η μουσική. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ λοιπόν, να δούμε πώς θα εκπαιδεύσουμε τους ε, επαγγελματίε σε αυτό το τρίτο σε αρχαιότητα επάγγελμα του κόσμου και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Λόπες, ε, πολύ ωραία, πώς θα βρούμε για τα ενιδρία τα κατάλληλα ψάρια. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εικόνα, γιατί τα ψάρια γνωρίζουν ε, εξορισμού να ε, κολυμπούν, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τα κατάλληλα ψάρια για το ενεδρίο μας. Και μην ξεχνάτε και αυτό το έγγραφο, το μικρό αυτό έγγραφο φυλάδιο. Ε, το Hints απαρτίζεται από τους επικεφαλείς των υπηρεσιών διερμηνίας όλου του κόσμου και έχουμε μια εφταετία που συναντιόμαστε. Βλέπετε ο χρόνος πραγματικά περνάει πολύ γρήγορα και αυτό που ενδιαφέρει τη Χίντς είναι πού θα περάσει τη σκητάλη, τι θα γίνει με την επόμενη γενιά, πώς θα βοηθήσουν οι οργανώσεις και οι αρμόδιοι φορείς για τη σωστή εκπαίδευση των διερμηνέων. Βλέπετε είναι σε τέσσερις γλώσσες, βλέπετε τις υπογραφές των μελών του Χίντς και θα καταλάβετε από το έγγραφο αυτό τι ψάχνουμε από, και τι περιμένουμε από τους εταίρους μας, από τα πανεπιστήμια για να υλοποιήσουμε το σκοπό μας. Γιατί η διερμηνία είναι ένα μείγμα τέχνης και επιστήμης. Εδώ δεν θα ασχολούμαστε με το επιστημονικό τμήμα, αλλά είναι και μια τέχνη διερμηνία και θέλουμε να, βρούμε την, να αναδείξουμε την αξία της και να ε, συνδυάσουμε το θεωρητικό και το πρακτικό σκέλος. Και όπως συμβαίνει και με την ιατρική και με την νομική επιστήμη, προσπαθούμε να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας και να βρούμε έναν τρόπο επιμόρφωσης ε, και μαθητείας που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα ενισχύσουμε και τις δικές μας προσπάθειες αλλά και θα βρούμε και εμείς ε, τους σωστούς επαγγελματίες που χρειαζόμαστε και που δυστυχώς σπανίζουν αυτή τη στιγμή. Οι συναδελφοί μου θα μιλήσουν για τα προβλήματα που έχουμε στην αναζήτηση ενός ε, οικονομικά βιώσιμου προγράμματος στα κοινωτικά θεσμικά όργανα για το θέμα αυτό Επίσης πώς θα ξεπεράσουμε τα γλωσσάρια και την τεχνολογία και όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας το πρωί ή μάλλον ε, η Επίτροπος Βασιλείου είπε το πρωί ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την διδασκαλία των γλωσσών, ούτε θα μετατρέψει τους κακούς δασκάλους ε, ε, σε καλούς, ούτε έναν αδιάφορο μαθητή σε γλωσσική διάνοια. Οι νέες τεχνολογίες είναι απλώς ένα εργαλείο. Θα πρέπει όμως να βρούμε κάποιον που δεν θα είναι μόνο ένας άνθρωπος που θα γίνει γέφυρα μεταξύ των πολιτισμών όπως μας είπε ο κύριος Λόπες αλλά θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται ε, και τις ιδέες, γιατί δεν μπορούμε να εντάξουμε σε κάποιον να σκέφτεται, αλλά θέλουμε και αυτό το χαρακτηριστικό από ένα διερμηνέα. Θέλουμε έναν επαγγελματία που άσχετα από τις γλώσσες που έχει ε, μάθει θα πρέπει να μιλάει καταπληκτικά την μητρική του γλώσσα και αυτό είναι δυσέβρετο τη σήμερα ημέρα, φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Επίσης ε, θα πρέπει να μπορεί να είναι και αγορητής να αγορεύει δημόσια και για την επακολουθητική και την ταυτόχρονη διερμηνία. Θα πρέπει να μπορεί να συγκεντρώνει και να συνδέει πληθώρα πληροφοριών και επίσης θα πρέπει να έχει και μια συνήθιστη και σπάνια μνήμη για θεσμικά θέματα. και επίσης θα πρέπει να τρώει σαπουλάκι, να πηγαίνει σπανίως στην τουαλέτα. Είναι δύσκολα αυτά. Πού να βρει κανείς καλό διερμηνέα που να έχει τόσα προσόντα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Σάλι Μπέιλι. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Η Όλγα Κοσμίδου μας ε, έβαλε ένα στίχημα το οποίο θα πρέπει όλοι, στο οποίο θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε, να ενισχύσουμε δηλαδή τη συνεργασία και να δουλέψουμε, να, να δικτυωθούμε. Και θα έλεγα ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η εμπιστοσύνη εγώ θα ήθελα απόψε να σας μιλήσω για κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε εταιρική σχέση στο μέλλον ανάμεσα στις σχολές διερμηνίας και τους επικεφαλείς ε, διερμηνείς ε, των διεθνών οργανισμών. Πρόκειται, είναι ένα θέμα εμπιστοσύνης. Όλοι έχουμε τη δουλειά μας. Εγώ δεν θέλω να κάνω τη δικιά σας δουλειά που είναι να ε, φτιάξετε καινούργιε διερμηνεί και δεν πιστεύω πω μπορείτε κι εσεί να κάνετε τη δική μου δουλειά, δηλαδή να προσφέρετε σε ένα διεθνή οργανισμό διερμηνή ποιότητα μέσα σε πολύ διαφορετικέ συνθήκε. Ε, Όμω, ακόμα και αν ο καθένα από εμά κάνουμε τη δουλειά μα και αν δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε επαγγέλματα, ο ένα εξαρτάται από τον άλλον. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε εσά για να μου δώσετε το υλικό που χρειάζομαι για να κάνω τη δουλειά μου και εσεί χρειάζεστε εμένα ώστε να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα προϊόντα που εσείς κατασκευάζετε, αν μπορώ έτσι να χαρακτηρίσω τους διερμηνείς, αλλά και εγώ διερμηνέας είμαι, οπότε μην ε, σας πειράξει, ε, για να μπορέσω να λανσάρω το προϊόν σας λοιπόν στην αγορά. Και αν εγώ δεν λανσάρω το προϊόν σας στην αγορά, δεν μπορείτε να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και αντιστρόφως ανάλογα Πρέπει να σας πω ότι αυτό το συνειδητοποίησα, διότι η δραστηριότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εξελιχθεί. Ε, για χρόνια ήμασταν ένα αριθμιστικό όργανο. Έχουμε φτιάξει 200 συμβάσεις ε, σε 40 και πάνω χρόνια. Όλα αυτά γίνονταν ε, σε δύο γλώσσες, στην έδρα, με προσλήψεις σε χώρες όπου υπήρχαν εξαιρετικές σχολές διερμηνίας. Δηλαδή θεωρούσαμε δεδομένη την ποιότητα των προϊόντων που φτάναν στην αγορά. Και έπειτα αυτή η δραστηριότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελίχθηκε μετατραπήκαμε, μεταμορφωθήκαμε σε ένα όργανο συνεργασίας, τεχνικής βοήθειας, έναν οργανισμό που πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα που εμείς είχαμε εκπονήσει όντως εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και τελείως άλλαξε η δραστηριότητα του Διερμηνέα που αντί για Διερμηνέα στην έδρα αγγλογαλλικά ε, μετατράπησε διερμηνέα περισσότερο σε consecutive με τις επίσημες γλώσσες που είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά και τι τις γλώσσες των χωρών μελών μας και χρειάστηκε να πάω για ψώνια σε μια αγορά τελείως διαφορετική όπου δεν είχα σχέση με φημισμένες σχολές διερμηνίας γνωστέ. και χρειάστηκε να φτιάξω, να χτίσω ε, σχέσεις εμπιστοσύνη για να δω αν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στι σχολέ αυτέ. Και εκεί ακριβώς οι εκπρόσωποι που είστε εσείς σχολών που είναι λιγότερο γνωστός, που έχουν λιγότερη εμπειρία, όπου ε, η εμπιστοσύνη πρέπει να δημιουργηθεί, είχα να κάνω πολύ δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, να, εμπνεύσουμε, να εμπνεύσετε εμπιστοσύνη στον ε, αρμόδιο για την πρόσληψη διερμηνέων οι ίδιοι οι δάσκαλοι ε, θα πρέπει να είναι διερμηνεί. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Ε, δεν μπορεί κανείς να διδάξει ένα επάγγελμα το οποίο είναι ένα επάγγελμα ειδικό, το οποίο το καταλαβαίνουμε μόνο όταν έχουμε εμεί οι ίδιοι ανάψει το μικρόφωνο και έχουμε αισθανθεί οι ίδιοι την αδρεναλίνη που περνά από τι φλέβε μα. Μόνο όταν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει ακριβώ αυτό και σε ποιο βαθμό απαιτεί την κινητοποίηση τη συγκέντρωση και των πόρων που έχει ο καθένα μα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οι σχολές που δεν το έχουν καταλάβει αυτό δεν μπορούν να μου δώσουν δυστυχώ το υλικό που χρειάζομαι για να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα. Δηλαδή, σχολές που έχουν καθηγητές που είναι διερμηνείς και που άρα επειδή ακριβώ είναι οι ίδιοι διερμηνεί, δεν θα φοβηθούν να μην δώσουν ένα πτυχίο αν ο υποψήφιο δεν το αξίζει. Και αυτό είναι, είναι ε, το, το θεμέλιο. Πρέπει δηλαδή να μπορεί κανεί σε ένα χρόνο να μην φτιάξει διερμηνεί. Είναι ο μόνο τρόπο για να μπορεί να έχει σε ανα πάσα στιγμή την εγγύηση να έχω εγώ την εγγύηση ότι όσοι έχουν το πτυχίο, στο πτυχίο του το όνομα της σχολής σας, γιατί αυτό κάνετε στην ουσία, δίνετε σε αυτούς τους ερμηνείς μια κάρτα, ένα επισκεπτήριο. Και όταν το βλέπω αυτό να μπορώ να τους προσλάβω με κλειστά τα μάτια. Να μπορείτε δηλαδή να μην δώσετε το πτυχίο αν δεν το αξίζει ο δερμηνέας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για τη σκητάλη, για το γεγονός ότι μας λείπουν διερμηνείς όσο πάει και περισσότερο. Είναι όντως ότι είναι πρόκληση η αλλαγή βάρδιας αυτή, αλλά η ανάγκη ε, για διερμηνείς δεν θα πρέπει σε καμία στιγμή να μας κάνει να αφινταλαντευόμαστε όσον αφορά την ποιότητα. Και αυτή η οργαν... αυτός ο οργανισμός που είναι πολύ πιο μικρός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται όμως διερμηνής και υποφέρει από το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετούς διερμηνείς για δεύτερη βάρη στην ουσία παίρνει διερμηνείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή δηλαδή που κάποιο κράτος μέλος αποκτά το καθεστώς ε, ειδική σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γίνεται υποψήφια χώρα είτε ούτως ή άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία παίρνει από την αγορά όλους τους διερμηνείς, τους ε, στραγγίζει είτε ε, απασχολώντας τους από τη χώρα τους, είτε καλώντας τους εδώ στις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν αδειάζει η αγορά, αδειάζει η αγορά στην λόγο χώρα. Εκεί που εγώ τους χρειάζομαι. Πρέπει πάντοτε να φτιάχνονται καινούργιοι διερμηνείς ποιότητας, αλλά και διερμηνείς που να μείνουν στη χώρα τους, στη χώρα προέλευσής τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν μικρό οργανισμό όπως ο δικός μου. Και επαναρχόμαστε διαρκώς σε αυτό το ίδιο ερώτημα που είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που ήθελα να σας διαβιβάζω και δίνω και πάλι το λόγο στην Κλέρ που θα έχει να πει άλλα πράγματα φαντάζομαι. Actually, I don't have other... Well, I don't have something different to say. I... Δεν έχω να πω τίποτα διαφορετικό. Συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε η Σάλη. Θα προσπαθήσω να πω διαφορετικά. Ενδιαφέρον αυτό που είπες για τη δυναμική που αλλάζει στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως προς τις γλώσσες. Και το βρήκα και πολύ ενθαρρυντικό από την ομιλία του κυρίου Λόπης, τη δυναμική, πώς αλλάζει, τη σχετική δυναμική και δύναμη των διαφόρων γλωσσών και όσα βλέπει να αλλάζει αυτή η δυναμική. Οι δύο επίσημες γλώσσες, όπως και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι αγγλικά και γαλλικά. Και θα σκεφτόταν κανείς ενδεχομένω ότι σιγά σιγά θα εξαφανιστεί η διερμηνία από τον όσα. Κάποια στιγμή όμως φάνηκε ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε de facto και ότι διατηρούσαν τη διερμηνία ως φιλοσική, ας πούμε, επειδή τα γαλλικά ήταν επίσημη γλώσσα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια μετακίνηση τεκτονικών πλακών. Το αγγλοαμερικανικό μοντέλο, με λίγους Γάλλους που αντιστέκονται, έχει αλλάξει. Και έρχεται σε πρόσκρουση με την γαλλόφωνη Αφρική και την ισπανόφωνη Φίλιο. διότι έχουμε περισσότερη συνεργασία με την παγκοσμιοποίηση, και ευρύτερη. Υπάρχει μια μετατόπιση λοιπόν και αλλαγή στη συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των διαφόρων γλωσσών και όλο και περισσότερο ε, καλούμαστε να ε, προσλαμβάνουμε διερμηνείς από άλλες γλώσσες ρωσικά και ισπανικά κυρίως αλλά και αραβικά, ε, ιταλικά, κινέζικα, ιαπωνικά και λιγότερο γερμανικά. Δηλαδή μετατοπίζεται εδώ η δυναμική και πάλι. Τώρα, στον θεωρούμε πολύ σημαντικό να διαδραματίζουμε ένα ενεργό ρόλο στην ένταξη ε, προσφάτως ε, αποφυτισάντων επιτυχιούχων. Είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ε, προσέλκυση των διερμηνέων, αλλά διερμηνείς που μόλις έχουν αποφοιτήσει είναι πάρα πολύ ε, καλή, είναι άριστη, ε, ενθουσιώδης, ε, συνειδητοποιημένη, ευσυνείδητη και ειλικρινά χαίρονται στις συνεδριάσεις. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει πάντα, όταν έχει περάσει 40 χρόνια σε μια καμπίνα στη συνέχεια. Ε, βεβαίως, ε, και από τους 16 μονίμους υπαλλήλους μας τουλάχιστον οι 12 ε, πηγαίνουν ε, στις εξετάσεις, ε, δύο σχολές κυρίως του Παρισιού, στις δύο. Αν μας καλέσουν και αλλού πηγαίνουμε. Επίσης, αν θέλετε να κάνουμε διασκέψεις, διαλέξεις, επίσης δεχόμαστε και διερμηνείς ασκούμενους που κάνουν βοβή καμπίνα και εκπαιδεύουμε κιόλας. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστεύομαι λιγότερο από τις άλλοι είμαι πιο καχύποπτη. Δεν θα βάζα μέσω στην καμπίνα ε, ε που μόλις έχουν αποφυτίσει, αν δεν τους έχω ακούσει, στην τάξη, στο μάθημα ή στις εξετάσεις. Ανεξάρτητα από τη σχολή που έχουν βγάλει, ε, τους καλώ να δουλέψουν σε βουβή καμπίνα, τους ακούω και τους λέω τη γνώμη μου. Και μετά αποφασίζω αν θα τους προσλάβω ή όχι. Και μπορούν να επανέρχονται να κάνουν βουβή καμπίνα όσο θέλουν. Ε, γιατί είναι πραγματικά άριστοι, εξαιρετικοί πολλοί από αυτούς, αλλά και πολλοί άλλοι δεν είναι και ορισμένοι απλούστατα δεν είναι έτοιμοι. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα, μπορεί να είναι για τους ίδιους, διότι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα της αποφύτησης ε, από τη μια ε, και να βρουν αρκετή δουλειά για να μπορέσουν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Για μένα δεν είναι πρόβλημα γιατί τους ενθαρρύνω να κάνουν βοβή καμπίνα, άσκηση, ζητώ και από διερμηνείς ε, πεπειραμένους να τους βοηθήσουν, να τους παρακολουθούν και να τους συνοδεύουν και τελικά προσλαμβάνουμε. Όταν λέω ότι δεν είναι έτοιμοι, τι εννοώ. Η τεχνική τους μπορεί να μην είναι αρκετά καλή, μπορεί να έχουν προβλήματα κατανόησης ε, στα αγγλικά, ιδιαίτερα και σε άλλες γλώσσες κάποιων προφορών ή κάποιων ε, ομιλητών. Ορισμένοι από αυτούς δεν θα είναι ποτέ έτοιμοι για τον εξή λόγο. Ότι δεν έχουν καν τις βασικές ικανότητες και η βασική ικανότητα για μένα είναι να μπορεί κανείς να μεταδίδει ένα μήνυμα με τρόπο αξιόπιστο σε ένα άλλο ακροατήριο. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα ακαδημαϊκά και πολύ βαριά δηλαδή και επικεντρώνονται στην τελική ε, ε, τεχνική εκπαίδευση, στη διαδικασία, κάνουν πάρα πολύ ε, ταυτόχρονη διερμηνία και πρακτική με διάφορους τρόπους, αλλά στερούνται των βασικών εφοδίων οι φοιτητέ. Και αν δεν τα έχουν βγαίνοντα από τη σχολή, αυτό δεν είναι κάτι που θα αποκτηθεί. Μπορεί να βελτιωθεί η γλώσσα, μπορεί να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη που έχουν και η εφράδειά τους, αλλά τα βασικά δεν πρόκειται να τα αποκτήσουν εκτός σχολής. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Βεβαίως με χαρά να συνεργαστούμε για να το μεταδώσουμε. Αν είναι και άλλοι έτοιμοι να τα ακούσουν, να συμφωνήσουν και να μοιραστούν μαζί μας αυτό το μήνυμα. Και με μεγάλη χαρά να προσλάβουμε για όλους αυτούς τους λόγους ε, πρόσφατα πρόσφατους πτυχιούχους και όλους τους λόγους που είναι βασικά εγωιστικοί. Ελπίζω να έχουμε κάποια τροφή για σκέψη για να έχουμε μια ζωηρή συζήτηση. Κανονικά μέχρι τις 6.30 είχε προβλεφθεί η διερμηνία, αλλά ελπίζω να παραταθεί λίγο το, το ωράριο των διερμηνέων, αν δεν έχουν αντίρρηση. Θα ήθελα να ακούσω και λίγα μαλτέζικα, γίνεται. Υπάρχουν ερωτήσεις. Χάρη, παρακαλώ το όνομά σου και από ποιο θεσμικό όργανο. Από το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σανγκάη. Και μάλιστα θα θέσω την ερώτησή μου την μητρική μου γλώσσα, τα κινέζικα και έχω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους την αγγλική και τη γαλλική καμπίνα που θα με μεταφράσουν. Η ερώτησή μου είναι απλούστατη. Το Πανεπιστήμιο μας της Αγκάης, από τότε που ξεκίνησε, που πρωτοξεκίνησε, έχει εκπαιδεύσει για 8 χρόνια διερμηνή συνεδρίων, πληρώντας τις διεθνείς προδιαγραφές για τους αποφύτους. Οι πτυχιούχοι μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διερμηνία. Επειδή όμως είναι Κινέζοι υπήκοοι, ε, έχουν ίσως πρόβλημα γιατί θέλουν πολύ ευχαρίστω να προσληφθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι βέβαια να, γίνει, να γίνουν τα κινέζικα επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν δυνατότητα να προσληφθούν ως μόνιμο προσωπικό, μόνο σε θέση freelance μπορούν να προσβλέπουν. Και Ε, φυσικά, επειδή είναι και γεγραμμένοι μέλη τη, ΑΕΚ, δεν μπορούν να ισχυριστούν ψευδώ ότι η έδρα του είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που κατάγονται από την Κίνα και ζουν στην Κίνα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αρκετά κονδύλια για να τους πληρώσει εισιτήρια business για να έρθουν να εργαστούν από την Κίνα στις Βρυξέλλες. Βέβαια, πιστεύω ότι ικανοί και καλή διερμηνείς μπορεί να έρχονται και από την Κίνα για να δουλεύουν στα κοινωτικά θεσμικά όργανα, αλλά δυστυχώ κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο για πρακτικούς λόγους. Ερωτώ λοιπόν, μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνουν ειδικέ θεωρήσεις στους διερμηνείς αυτούς, ώστε να μπορούν να έρχονται ε, να σπουδάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εργάζονται και ως freelance στα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, Χάρη. Θα ήθελα κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στο Χάρη. Κύριε Χιμένες Μαρίνη, πως εσείς και παρακαλώ οι απαντήσεις να είναι όσο πιο λακωνικές γίνεται για να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις προλάβουμε. Καταρχήν χάρη, όντως ε, ισχύει ο κανόνας ε, που επιτρέπει μόνο μία επαγγελματική έδρα. Δεν μπορεί κανείς να έχει ταυτόχρονα δύο επαγγελματικές έδρες. Βέβαια, είναι δυνατό ένας Κινέζος διερμηνέας να κάνει μελέτη της αγοράς εργασίας στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφασίσει να μεταφέρει την έδρα του για ένα εξάμεινο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου να εργαστεί κυρίως για θεσμικά όργανα που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και το δεύτερο, το άλλο εξάμεινο να εργάζεται στην Κίνα. Αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα ούτε είναι κάτι άγνωστο, γιατί πολλοί διερμηνείς ακόμη και κοινοτικών γλωσσών το κάνουν συστηματικά. Συστηματικά αλλάζουν την έδρα τους. Και μάλιστα και οι διερμηνείς των Ηνωμένων Εθνών τακτικά εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, γιατί θέλουν να συνδυάσουν την ιδιωτική αγορά αφενός με μια πιο θεσμική αγορά ή με την αγορά των διεθνών οργανώσεων ή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Έτσι θα μπορούσε ένα Κινέζο να εργαστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση πάντω του δικού μα κανόνε, γιατί μα δεσμεύει η συλλογική σύμβαση που έχουμε συνάψει με τους ε, freelance διερμηνείς ε, προβλέπει ότι για τους ε, διερμηνείς που δεν έχουν έδρα τις Βρυξέλλες τους πληρώνουμε το αεροπορικό εισιτήριο υπό όρους όμως το εισιτήριο θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι ενός αθέμητου ανταγωνισμού παροτρύνοντας διερμηνείς να εργάζονται σε συνθήκες που αντιβαίνουν στα φυσικά τους δικαιώματα. Ευχαριστώ, Χουαν Κάρλος. Ερώτηση από το πίσω μέρος σας. Ευχαριστώ. Βίτος Γκαβρόσκι, είμαι μέλος της ΑΕΚ και μάλιστα εκπαιδεύω διερμηνείς στο Πανεπιστήμιο του Ποσνάν στην Πολωνία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μας είπε η κυρία Όλγα Κοσμίδου και η κυρία Σάλι Μπέιλι. Μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δύο γιατί πραγματικά είχαν πολύ σημαντικά σημεία που αφορούν άμεσα όχι μόνο εμάς τους διερμηνείς αλλά και τους Πριτάνης που συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη. Δηλαδή, θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο αλήθειες που είναι γνωστές αλλά καλό θα ήταν να τις επαναλάβουμε. Η πρώτη αλήθεια είναι η απάντηση στην ερώτηση. Ποιος θα πρέπει να ε, ε, ε, επιμορφώνει τους διερμηνείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι επαγγελματίες διερμηνείς που έχουν διδακτικές ικανότητες. Ποιος δεν μπορεί όμως να εκπαιδεύει διερμηνείς. Και αυτό το βλέπουμε συχνά στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να διδάσκουν και να επιμορφώνουν διερμηνείς άνθρωποι που δεν είναι διερμηνείς επαγγελματίες. Για παράδειγμα, μερικές φορές είναι εκπρόσωποι φιλολογικών σχολών, είναι φιλόλογοι. Μπορούν να διδάσκουν αυστριακή λογοτεχνία για παράδειγμα και αυτοί ε, εκπαιδεύουν διερμήνες. Κατά τη γνώμη μου είναι ακατάλληλοι τέτοιοι άνθρωποι για την εκπαίδευση διερμήνων, δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι οι ίδιοι επαγγελματίες διερμηνείς. Και έχω και μία έκκληση. Εδώ και 21 χρόνια ε, είμαι επικεφαλής της ε, Σχολής Διερμηνίας ε, στο Πόσναν και έχω στερές επαφές με τους Πριτάνης και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση και να παροτρύνω τους Πριτάνης αν υπάρχουν τέτοια είδους τμήματα και διαμορφωθούν και στελέχη για την διδασκαλία αυτή, θα ήθελα αυτές οι, αυτά τα τμήματα να ε, εξαρτώνται, να υπάρχονται άμεσα στους Πριτάνης. Γιατί όπως είπε ο καθηγητής Λέντερ σε μία διάλεξη, η διερμηνία συνεδρίων δεν έχει και πολλά κοινά στοιχεία με τις γλώσσες μερικές φορές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ, πολύ. Θα ζητήσω από την Όλγα Κοσμίδου να σχολιάσει και μετά την Κλέρ ε, Ντόναβαν να προσθέσει τις παρατηρήσεις της. Νομίζω πως το είχα ήδη πει στη διάρκεια της παρέμβασής μου ότι και καταρχήν αναφέρθηκε και η δήλωση Hints που βρίσκεται σε όλους τους φακέλους και σας ε, παροτρύνω να τη διαβάσετε. Το, και νομίζω πως το είπα και στην παρέμβασή μου ότι ούτε οι φιλόλογοι ούτε οι καθηγητές γλωσσών μπορούν να διδάξουν την ε, διερμηνία. Ε, είναι κάτι το οποίο με εκπλήσει και με λυπεί Ότι δηλαδή θα μπορούσε κάποιος πρίτανης να ζητήσει από κάποιον που δεν είναι γιατρός να διδάξει την ιατρική. Ποτέ δεν θα σκεφτόταν ένας πρίτανης να επιτρέψει σε κάποιον που δεν είναι ε, νομικός να διδάξει το ε, νομική. Δεν καταλαβαίνω τι σου μαγικό γίνεται και να, ώστε να πιστεύει πως ένας πολύ καλός φιλόλογος μπορεί να ε, διδάξει την διερμηνία. Η Χίντς, η επικεφαλή δηλαδή των ε, διαφόρων βημάτων διερμηνίας σε διεθνεί οργανισμούς, είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Και η Κομισιόν έχει πολύ πιο ξεκάθαρη θέση, πιο σκληρή θέση, ότι δεν συνεργαζόμαστε παρά μόνο με τι σχολέ που όχι μόνο δεν απασχολούν παρά μόνο διερμηνείς, αλλά μάλιστα διερμηνείς οι οποίοι είναι διαπιστωμένοι από κάποιον μεγάλο διεθνή ε, οργανισμό. να μην απαιτούν από τους διερμηνείς να έχουν διδακτορικό πτυχίο, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες διερμηνείς και που έχουν ε, διδακτορικό στην κατοχή τους. Μάλιστα, δύο-τρεις από αυτούς βρίσκονται εδώ στην αίθουσα είναι παρόντες. Λοιπόν, δεν πρέπει να πετούν διδακτορικό, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να ε, διώχνουν τους διερμηνείς και να μην απαιτούν από τους ε, διδάσκοντες να μην εργάζονται πια. Λέγοντας, ναι, τώρα είστε υπάλληλοι του Πανεπιστημίου ή κρατικοί υπάλληλοι και άρα δεν μπορείτε να εργαστείτε ως διερμηνείς. Κανένας γιατρός δεν θα το δεχόταν αυτό. Κανένας γιατρός δεν το δεχόταν αυτό. Και είναι κατανοητό γιατί δεν θα ήξερε πια ποια είναι οι νέες εξελίξεις, νέες μέθοδοι ιατρικής. Οι νέες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη του. Γιατί ένας ε, διερμηνέας να κοπεί, αποκοπεί από την καθημερινή του δουλειά και να συνεχίσει να διδάσκει τα όσα γίνονταν τον προηγούμενο αιώνα. Μα με ποια λογική μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορεί ένας πρίτανας να το σκεφτεί αυτό. Γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει και καλέσαμε εδώ τις πανεπιστημιακές αρχές για να τους πούμε ακριβώς ότι πρέπει ότι μάλλον βλάπτουν τη φήμη των πανεπιστημίων τους εάν κάνουν τέτοιο είδους πρακτικές. Είναι είναι, είναι πολύ σημαντικό όποιος διδάσκει τη διερμηνία να είναι διερμηνέας και να συνεχίζει κιόλας ε, να ασκεί το επάγγελμά του. Um, very much along the lines of what Olga's already said. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με το όσα είπε η Όλγα ήδη, αλλά είπατε ότι συμφωνείτε και ότι η αλήθεια είναι ότι ένας ε, διερμηνέα που επαγγελματίας θα πρέπει να διδάσκει διερμηνία και όχι άλλοι και σε αυτό συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας πραγματικός ορισμός του διερμηνέα και Γι' αυτό και δίνει αυτό το πιο αυστηρό ορισμό το Ευρωκοινοβούλιο, πράγμα που είναι κάπως αντιφατικό. Το πρόβλημα είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι είναι διερμηνέας, αν τύχει που και που να κάνει λίγη διερμηνία. Και αυτό συμβαίνει τακτικά σε διάφορα μέρη του κόσμου που έχω επισκεφθεί. Ότι δηλαδή κοσμο που είναι δάσκαλοι γλωσσών, α πούμε, κάνουν και που και που λίγη διερμηνία και λένε ναι, είμαι διερμηνέα δεν είναι ότι θα πρέπει απλά να, είναι διερμηνείς, αλλά είναι και καλοί διερμηνείς, ώστε σωστά να μπορούν να διαβάσουν τις δεξιότητές τους. Μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να είναι κάπως αντιφατικό το να επιμένουμε και να λέμε ότι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σε κάποιον οργανισμό, γιατί ίσως σε ορισμένες αγορές να μην υπάρχει τέτοιο οργανισμό και η γλώσσα τους να μην χρησιμοποιείται από διεθνείς μεγάλους οργανισμούς. Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι μια καλή βάση να είναι μέλη της ΑΕΚ για παράδειγμα. Και αυτό βοηθάει να διευκρινιστεί κάπως ε, για το για ποιον μιλάμε. Εμείς και εσείς λοιπόν, εσείς ως εκπαιδευτές και εμείς ως ε, εργοδότες και εγώ είμαι ψυχολογικά ε, λίγο και από τα δύο έχουμε τεράστια ευθύνη όσον αφορά την πολυγλωσία διότι ο κύριος Λόπες είπε ότι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τον διερμηνέα, να εμπιστεύεται τον διερμηνέα και το μήνυμα που περνάει. Και αυτό μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα μόνο όταν δει ο άλλος ότι η διερμηνέα είναι καλή. Αν εμείς προσλαμβάνουμε κόσμο που δεν είναι καλός, γιατί είναι πιο βολικό, φθηνότερο, γιατί δεν ζουν πιο κοντά κτλ. για οποιοδήποτε λόγο, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγηση, αν τους εκπαιδεύουμε, τους δίνουμε ένα πτυχίο, ενώ δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες ενό διερμηνέας, τότε στην ουσία βάζουμε αυτό γκολ και πραγματικά δεν εξυπηρετούμε καθόλου την πολυγλωσία. Barbara. Barbara. Και θα είναι τα τελευταία ερώτηση, μου λέγουν. Δεν είναι ερώτηση, ένα σύντομο σχόλιο, η κυρία Μόζερ ε, Μέρσερ. Αφού μιλούμε για πρότυπα, θα ήθελα να πω ότι Έχουμε ένα νέο έγγραφο για τα πρότυπα ποιότητας για όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης διερμηνέων και ίσως με μεγάλη χαρά να μπορώ να σας πω ότι ε, από σήμερα ο Όμιλος, αυτό το κονσόρσιουμ ε, είναι έτοιμος, έχει ανοίξει για τις υπογραφές και μπορείτε τα διάφορα πανεπιστήμια που ενδιαφέρεστε και θέλετε να γίνετε μέλη και είναι πολλά να το συμβουλευτείτε στο διαδίκτυο. Πάντως πολλά από όσα υπόθηκαν συμπεριλαμβάνονται ε, σε αυτά τα στάνταρ και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Ήθελα μόνο να το αναφέρω. So I you all of you. Σας ευχαριστώ όλους σας, κύριε Κοσμίδου. Θα ήθελα να χειροκροτήσετε τους διερμηνείς μας. and let's proceed for our Μια οργανωτική παρατήρηση. Ζητώ συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Ε, την υπομονή σας. Ευχαριστώ τη Βάτση και όλους τους άλλους. Ε, πάμε τώρα στη δεξίωση και στο δείπνο. Ε, θα σας συνοδεύσουν οι αγαπητοί μας ενεργάτες και βοηθοί. Όσοι δεν μπορείτε να έρθετε τώρα... Ε, ή στο δείπνο ε, στις 9.30 ώρα ακριβώς αρχίζουμε αύριο το πρωί χωρίς ακαδημαϊκά τέταρτα και πολύ συχνά υπάρχουν ουρές στον έλεγχο ασφαλείας, οπότε καλό θα ήταν κατά τις 9 να είστε εδώ και να έχετε μαζί σας και το θαυμάσιο μπάτζ, την κάρτα εισόδου. Και ένα τελευταίο, ελπίζω να έρθουν και οι διερμηνείς, παρόλο που αύριο το πρωί... Ε, ε, θα ακούσουμε για το πόσο καλά μπορούν να μεταφράζουν οι αυτόματες μηχανές. Αλλά να έρθουν και οι συνάδελφοι να δουλέψουν. Ε, ευχαριστώ.